Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Να σας ε, ευχηθώ κι εγώ γιατί είναι η πρώτη φορά που συνεδριάζουμε στο νέο έτος. Ελπίζω να είναι αποδοτικές οι εργασίες μας. Πρέπει καταρχάς να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Έχετε αντιρρήσει, μήπω κύριε Γιάρ, για την ημερήσια διάταξη. Όχι, ωραία. Δεύτερο σημείο. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 11ης και 12ης Νοεμβρίου 2019 και Δευτέρας και 3ης Δεκεμβρίου 2019. Έχουν διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής τα πρακτικά. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αντίρρηση. Εφόσον δεν υπάρξει κάποια ένσταση, θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Και προχωρούμε. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Σας ενημερώνω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ως προς τα ακόλουθα σημεία. Έχουμε τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας ε, για τα σημεία B, Β, στις 11-12 Νοεμβρίου του 2019, που είναι τα εξής σε ό,τι αφορά τις αναφορές 646 του 2018, 755 του 2018 και 145 του 2019 παραμένουν ανοιχτές και θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη μιας προσεχούς συνεδρίασης. Εν συνεχεία έχουμε την αναφορά 171 του 2019, η οποία διατηρείται και αυτή ανοιχτή και θα περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη προσεχού συνεδρίασης και θα σταλεί προ ενημέρωση και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ΕΝΒΗ. Έχουμε μετά τις ε, εξή δύο αναφορές, 145 του 2019 και 211 του 2019. Για τι εν λόγω αναφορές, οι αναφέροντες ε, θα έχουν διορία δύο μηνών για να αντιδράσουν μετά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επόμενη αναφορά, η υπαριθμόν 690 του 2018. Παραμένει ανοιχτή και θα την εξετάσουμε από κοινού με την αναφορά 784 του 2019. Τώρα, οι αναφορές 124 του 2019 και 178 του 2019 κλείνουν. Σε ό,τι αφορά τι ε, φυσβητούμενε τάσει, έχουμε τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας. Εγκρίνονται οι συστάσεις ε, υπό τη μορφή που πρότεινε η για τις αναφορές. 505 του 2019, 515 έως 5.41 και 5.55 και μετά έχουμε τη 5.36, 5.51, 5.63, 5.96 όλες το 2019 που εγκρίνονται με βάση τα όσα πρότειναν οι πράσινοι. Αυτά σε ό,τι αφορά τις ε, ανακοινώσεις. Το λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη το σημείο αυτό και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε συζητήσεις ε, για τις διάφορες αναφορές. Καταρχάς έχουμε το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης ε, για αναφορές που άπτονται θεμάτων του ανταγωνισμού. Καταρχά, θα συζητήσουμε την αναφορά 984-2018 για τη διαδικασία για την πώληση των λιμπτοπαραγωγών μονάδων της ΔΕΗ ε, της Δημόσιας Επιχείρησης Ελεκτρισμού της Ελλάδος για τις ε, τοποθεσίες Μελίτη και Μεγαλόπολη. είχαμε ενημερωθεί για το ότι δεν θα είναι παρόν ο αναφέρον. Επομένω, το λόγο έχει ευθύ αμέσω ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φραντσέσκα Ματέρε, κάπω έτσι. Φραντσέσκο Ματέρια, ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα φορά φορά τις δεσμεύσεις που έχει προτείνει η Ελλάδα ε, το 2018 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί το θέμα το ανταγωνισμό όσον αφορά την προνομιούχα πρόσβαση στο λιγνίτη που χορηγείται από την Ελλάδα στη ΔΕΗ ε, και στην, ε, μονάδα, στην, ε, στην εταιρεία εκποίησης. Είναι αντίθετη με την απόφαση 2008-2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τελικά στήριξαν τα δικαστήρια του 2016. Οι δεσμεύσεις του 2018 που υιοθετήθηκαν μετά τις αποφάσεις του ΔΕΚ προέβλεπαν ότι θα έπρεπε να εκποιήσει δύο μονάδες, τη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη, ο αρμόδιος φορέας, μέσω ανοιχτού διαγωνισμού και διαφανού. Εκποιώντα λοιπόν τι μονάδες του Λιγνίτη, διασκεδάστηκαν οι συνεχεί Ευρωπαϊκές Επιτροπή, διότι οι ανταγωνιστές ε, του αρμόδιου δημόσιου φορέα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση ε, στι μονάδε και τα μέτρα ε, προέβλεπαν διάφορα μέτρα διαφύλαξη για να προστατευτούν τα συμφέροντα του διαρμοδίου οργανισμού. Μετά από το, μακρύ διαγωνισμό που επεκτάθη η εκποίηση παρατάθηκε πολλές φορές κατόπιν αιτήματο τη ε, ελληνική δημοκρατία και του αρμοδίου φορέα για την πώληση τον Ιούλιο του 2019. Οι μονάδε λιγνίτου δεν είχαν πωληθεί από τον νομό φορέα και η Ελλάδα δεν μπόρεσε να εφαρμόσει τα διεθνωτικά μέτρα του 18. Τι συνέβη έκτοτε. Ε, βασικά, έχουμε νέα κυβέρνηση που ανέλαβε τα καθήκοντα τον Ιούλιο του 2019 και αυτή η νέα κυβέρνηση υιοθέτησε το Δεκέμβριο πέρσι νέο σχέδιο για την ενέργεια και για το κλίμα, εθνικό σχέδιο. Ευπρόσδεκτο το σχέδιο αυτό για την ενέργεια και το κλίμα προβλέπει ότι οι περισσότερες μονάδες του Λιγνίτη μέχρι το 2023 ε, θα σταματήσουν να λειτουργούν. Λόγω τη τρέβλωση όμως μέσω του, της ΔΕΗ και του αρμόδιου φορέα για την πώληση, αυτή θα παραμένει η κατάσταση μέχρι να σταματήσει η χρήση του λιγνίτη στην ε, χώρα και υπέχει ε, υποχρέωση να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΔΕΚ Ελλάδα του 2016 και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλέσαμε την Ελλάδα να υποβάλει σχετικά διορθωτικά μέτρα χωρίς να συνεχίσει να έχει την προηγούμενη πορεία και η Ελλάδα επίσημα μας ενημέρωσε ότι προτίθεται, το ανακοίνωσε το Νοέμβριο του 2019, να υποβάλει αναθεωρημένες δεσμεύσεις και να κλείσει αυτή η υπόθεση και τεχνικά μέτρα προβλέπουν ότι μέχρι να εξαλειφθεί πλήρη χρήση του λιγνίτη στη χώρα, οι ανταγωνιστές του δημόσιου φορέα θα έχουν πρόσβαση στην παραγωγή ε, ηλεκτρικής ενέργειας από την ε, καύση του λιγνίτη. Ευχαριστώ. Και τώρα Σωστό. Ο κ. Βίντα θα μιλήσει. Εκ μέρους του ΕΛΚ συμφωνούμε με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί σωστή προσέγγιση. Να ακολουθήσει διαθρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση, πράσινη προσέγγιση και να μην χρησιμοποιεί το λιγνίτης μετά το 2028. Έτσι το παρόν θέμα γίνεται απειρχιωμένο, ξεπερασμένο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα σημαντικό θέμα. Αφορά το περιβάλλον και το, τα θέματα του ανταγωνισμού. Σημαντικά θέματα, τα περί ανταγωνισμού, όμως Πιστεύουμε ότι αυτή η αναφορά θα μπορούσε να κλείσει εφόσον η απάντηση της Ελλάδας και η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής α, θεωρούνται βήματα αποδεκτά. Ευχαριστώ κύριε Βίντσεν. Ο κύριος Νικόλ Αλαβάνος ζητά το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εντάξει. Επιτρέψτε μου σύντομα και χωρίς πολύ καθυστέρηση να εκφράσω την δική μα άποψη, την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε, ε, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από την εκτίμηση που κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν σε σχέση με αυτές τις δύο μονάδες τι οποίες συζητάμε στην παρούσα αναφορά, ε, καθώς ε, ήταν, να πω ότι ήταν μια αναφορά στην οποία εμεί ετηθήκαμε να παραμείνει ανοιχτή και να έρθει ξανά σε συζήτηση. Κατά την άποψή μα, δεν θα έπρεπε να εντάσσεται στο ζήτημα τη ε, ανταγωνιστικότητα. Μάλλον θα έπρεπε να εντάσσεται στο, στο, κάτω από το θέμα τη ενέργεια. Το θέμα για μα δεν είναι ε, το αν θα πουληθούν αυτέ οι μονάδε παραγωγή ηλεκτρικού ε, ρεύματο και σε τι τιμή. Το ζήτημα για μα είναι ότι δεν πρέπει να πουληθούν. Γιατί, αφενός γιατί είναι μονάδες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, έχουν χτιστεί την περίοδο που η ΔΕΗ ήταν δημόσια εταιρεία κοινού ωφέλεια, κρατική εταιρεία, με λεφτά δηλαδή του ελληνικού λαού, των Ελλήνων εργαζομένων, για να μπορούν να καλύπτεται οι ανάγκε των λαϊκών οικοκυριών, των εργαζομένων και τη βιομηχανία τη χώρα σε ηλεκτρική ενέργεια. Αντιλαμβανόμαστε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο αφού και οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά και η τωρινή, θα πω και πιο συγκεκριμένα, και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και συνολικά όλες οι κυβερνήσεις, εφάρμοσαν το πλαίσιο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα με τη λογική της απελευθέρωσης της ενέργειας, στη συνέχεια με την πράσινη ανάπτυξη και τώρα με το ευρωπαϊκό πράσινο deal και την απολιγνητοποίηση. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν την πώληση και τη, ταυτόχρονα την ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ και τα λοιπά σε σχέση με του ρήπου στερούνται λογική. Γιατί πέρα από τι μονάδε τη Μεγαλόπολη, η μονάδα για παράδειγμα τη Μελίτης είναι μια μονάδα τελευταία τεχνολογία με πολύ χαμηλού ρήπου. Ακόμη στερούνται λογική, γιατί σήμερα υπάρχει η δυνατότητα με συντεταγμένο τρόπο με ενιαίο κρατικό έλεγχο τη ενέργεια, να γίνουν οι αναγκαίε επενδύσει έτσι ώστε οι μονάδε παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη να αποδίδουν υψηλότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πολύ χαμηλότερους ρήπους. Σαν πρώτο στάδιο, πρώτο βήμα, το οποίο θα επιτρέψει να έχεις μια παραγωγή ηλεκτροενέργειας στη χώρα που θα καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες του ελληνικού λαού πρώτα και κύρια. Στον αντίποδα αυτού, η πολιτική που εφαρμόστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, που είναι σε αυτό το πλαίσιο που είπαμε και πριν, απελευθέρωση της ενέργειας, πράσινη ανάπτυξη, απολιγνητοποίηση, είχε πάρα πολύ βαριέ συνέπειε για τον ελληνικό λαό. Ποιε ήταν αυτέ. Πρώτον, τεράστια αύξηση στα οικιακά τιμολόγια του ρεύματο, τα οποία φορτώθηκαν με φόρου και επιφόρων για την πράσινη ανάπτυξη, έτσι ώστε να μπορούν να επιδοτηθούν οι ιδιωτικέ εταιρείε που μπήκαν στο ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Χειροτέρευση των εργασιακών συνδικών των εργαζομένων μέσα στην ίδια την εταιρεία, με ευέλικτε σχέσει, με πολλών τύπων συμβάσει, και τώρα με το τελευταίο βήμα της κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και με πρακτικά κατάργηση και τη κλαδικής σύμβασης την οποία είχαν πετύχει οι εργαζόμενοι εκεί με τον αγώνα τους. Τρίτον, κατάτμιση και ιδιωτικοποίηση της ενιαία ΔΕΗ με αποτέλεσμα τώρα να γίνεται ένας μεγάλος ανταγωνισμός ιδιωτικών εταιριών ποιος θα πάρει ποιο τμήμα της ΔΕΗ. 5.000 απολύσεις που προϋπολογίζει η, αυτή, η ίδια η εταιρεία, η οποία πλέον λειτουργεί με κριτήριο ιδιωτική οικονομία, σαν ιδιωτική εταιρεία, σαν αποτέλεσμα κλεισίματο μονάδων, πωλήσεων όχι μόνο των λιγνητικών σταθμών παραγωγή, αλλά πωλήσεων και των υδροελεκτρικών φραγμάτων, μικρών και μεγάλων και άλλων κομματιών του δικτύου. Και βεβαίω πράγμα το οποίο θα οδηγήσει στην ένταση τη ενεργειακή εξάρτηση τη χώρα. Όταν μιλά για παραγωγή ενέργειας από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι ένας φόρος τον οποίο η Ελλάδα δεν διαθέτει, άρα θα πρέπει να τον εισάγει. Αντίθετα, ο λιγνίτης υπάρχει μέσα στο υπέδαφο τη χώρα, δεν κοστίζει τίποτα η εξόριξή του και η χρήση του για την παραγωγή ενέργεια. Και βεβαίω το σχέδιο αυτό τη απολιγνητοποίηση θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο στου εργαζόμενου τη ίδια τη εταιρεία, αλλά συνολικά στι οικογένειε, στου κατοίκου των περιοχών κυρίω τη Δυτική Μακεδονία, όπου εξαρτώνται άμεσα ή έμεσα από την παραγωγή ενέργεια και δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Εμείς νομίζουμε ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο προσανατολισμός που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα της ενέργειας, η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δηλαδή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράγμα το οποίο το πληρώνει πάρα πολύ βαριά ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες εργαζόμενοι. Στη χώρα μας είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει κρυθεί. Διεξάγονται αυτή τη στιγμή πολλοί αγώνε κινητοποίησης των εργαζομένων των κατοίκων των περιοχών τις οποίε και εμεί στηρίζουμε, η άποψη δική μα είναι ότι χρειάζεται ένα ενιαίος κρατικό φορέα ενέργεια, ο οποίο θα μπορέσει αξιοποιώντας όλε τις, τους τρόπους παραγωγής της ενέργειας να στηρίξει την ανάγκη για φτηνή ηλεκτρική ενέργεια για, την, ε, για τους εργαζομένους για τα λαϊκά νοικοκυριά και να καλύπτει τις ανάγκες ε, για τη βιομηχανία της χώρας κάτω από ένα σύστημα κεντρικού ενιαίου σχεδιασμού επιστημονικού όλης της οικονομίας. Με αυτή την έννοια και ακριβώς επειδή είμαστε σε φάση όπου η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, πατώντα πάνω στα βήματα που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εντείνει την πάλη για να ανατραπεί το σύστημα, για να πουληθεί ή να ιδιωτικοποιηθεί, να γίνουν απολύσει. Πράγμα το οποίο ήταν, και κλείνω με αυτό, και αντικείμενο τη πρόσφατη αξιολόγηση τη Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα όργανα τη, που επέμεινε για άλλη μια φορά στην κατεύθυνση αυτή Νομίζουμε ότι πρέπει στο φω των νέων στοιχείων που έχουμε στα χέρια μα και των κινητοποιήσεων που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα μέσα στη χώρα να μην κλείσει η, ε, η συζήτηση για αυτή την αναφορά, να κρατηθεί ανοιχτή και να παρακολουθήσουμε τι εξελίξει. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Νικολάου για τους σοσιαλιστές πιστεύουμε ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι σαφής και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περαιτέρω έρευνα για το θέμα αυτό. Είναι εξαιρετικά πολιτικό ζήτημα. Έχουμε θέματα υποχρεωτικής ιδιωτικοποίησης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η αναφορά αυτή πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστούμε κύριε Αγίους. Για τους πράσινους δεν βλέπω κανέναν. Και εμείς έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για τον διαγωνισμό αυτό, καθώς ε, η Επιτροπή στην απάντησή της είπε ότι θα υπάρξει δίκαιη προσέγγιση με βάση την κατάσταση της αγοράς για τον διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση αυτή. Οι αναφέροντες ωστόσο θεωρούν και φαίνεται εύλογο ότι η πώληση των δύο αυτών μονάδων στη Μελίτη και την Μεγαλόπολη είναι πολύ, γίνεται σε πολύ χαμηλότερο τίμημα από την τιμή της αγοράς. Τι θα πει δίκαιη τιμή με βάση τους κανόνες της αγοράς για μια συγκεκριμένη επιχείρηση όταν έχουμε μόνο δύο μονάδες τέτοιες. Αυτή είναι η παρέμβασή μου υπομορφή ρητορικού ερωτήματος. Δεν θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην αγορά. Ο κ. Αρβανίτης. Σας ευχαριστώ από την ε, αλλά από την αριστερά κύριε πρόεδρε θα συμφωνήσω με τη δική σας εκτίμηση δηλαδή συμπλέομαι στη σκέψη και τη δική σας αλλά και της ομάδας των σοσιαλιστών προσθέτοντας μόνο ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έθεσε ο συνάδελφός μου ο κύριος ε, αλαβάνος Μιλάμε και για χιλιάδε θέσει εργασία που έχουν άμεση σχέση ουσιαστικά με τι τοπικέ κοινωνίε. 5.000 άνθρωποι και βεβαίω ο συνδυασμό των ανθρώπων αυτών και των οικογενειών με τη γενικότερη εικόνα τη παραγωγή. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να επιμείνουμε, να μείνει ανοιχτό και θα πρότεινα να πάει και στην ΕΜΠΛ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι. I think uh, uh, that η απόφαση μπορεί να είναι εξή. Παραμένει ανοιχτή η αναφορά. Ζητούμε από την Επιτροπή να μας ενημερώσει για την έκβαση της νέας διαδικασίας πώληση. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή η διαδικασία ξεκίνησε πέρυσι το Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω των εκλογών. Λόγω των εκλογών, συγγνώμη. Λοιπόν, ζητούμε ενημέρωση και επικαιροποίηση του θέματος από την Επιτροπή και να προτείνω να στείλουμε το θέμα και στην Επιτροπή Απασχόλησης προς ενημέρωση. Ωραία, ευχαριστούμε. No. from the EPP. Okay, thank you. let's examine this case. Ωραία, συνεχίζουμε την εξέταση του θέματος ελπίζοντας σε μια καλύτερη λύση. Επόμενο θέμα. Σημείο 5. Τρεις αναφορές. 620 του 2018 από έναν Έλληνα πολίτη με 43 υπογραφές για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής εξόρυξης στην Χαλκιδική στην Ελλάδα. Εξόρυξη αλλά περιβαλλοντική προσέγγιση. Αναφορά 917 του 2013 του κυρίου Σωτήριου Δαμόπουλου, Έλληνα πολίτη, για την εξόριξη χρυσού στις, στις σπουδιές της Χαλκιδικής και της, ε, την περιβαλλοντική ρήπανση που προκύπτει. Και αναφορά 1 του 2016 από τον Ισμαέλ Αντώνιο Λόπες Πέρες, Ισπανό πολίτη, εξ της ε, ανεξάρτητης περιβαλλοντικής οργάνωσης Πετών Λόμπο, για την αποψήλωση του, του δάσους που προκλήθηκε από την ε, το ρηχείο των σκουριών στη Χαλκιδική Ελλάδα. Για να μην υπάρξει σύγχυση. Πρόκειται για τρεις αναφορές για το ίδιο θέμα, τον ελληνικό χρυσό, ελληνική ε, θηγατρική του Καναδέ, της Καναδέης εταιρείας Eldorado Gold που ε, λειτουργεί σε τέσσερις, περιοχές, τέσσερις διαφορετικές περιοχές στη Χαλκιδική. Έχουμε τρεις ομιλητές, αν έχω καταλάβει καλά. Δύο εκπροσωπούν τους, τον πρώτο αναφέροντα. Πέντε λεπτά και οι δύο. Πέντε λεπτά για την, τον δεύτερο αναφέροντα. Ο κύριος Κυριάκος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Κωνσταντίνος Ευθυμίου. Μαζί έχετε πέντε λεπτά. Ποιο θα μιλήσει. Θα προσπαθήσω να πω αυτά που έχω, αυτά που έχω γράψει όσο γίνεται συντομότερα. Ε, θα αναφερθώ στη μη τήρηση κατά την άποψή μου από την εθνική νομοθεσία της χώρας μου της οδηγίας 9243 η οποία αφορά τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίων τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν σημαντικά περιοχές του δικτύου Natura 2000 ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 και 4 της Οδηγίας 9243. Το βασικό αποτέλεσμα συμπέρασμα αυτής της οδηγίας είναι ότι ένα σχέδιο δεν εγκρίνεται παρά μόνο όταν η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου. Το άρθρο 6 παράγραφος 3 προβλέπει μια ειδική διαδικασία δέουσας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εφαρμόζονται σε κάθε σχέδιο μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διατήρηση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατό να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο καθεαυτό ή από καινού με άλλα σχέδια. Δηλαδή η αποκαινουμε αλλα αυτή εφαρμόζεται σε σχέδια τα οποία πρώτον δεν έχουν σχέση με τη διαχείριση του τόπου και δεύτερον ενέχουν κινδύνους σημαντικών επιπτώσεων στον τόπο. Πώς εφαρμόζεται αυτή η οδηγία στην, ε, εθνική, στην, Ελλάδα, στην, πώς έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία. Το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας αυτής ενσωματώθηκε όχι επιτυχώς κατά την άποψη πολλών νομικών στο εθνικό δίκαιο με μια κοινή υπουργική απόφαση και συμπληρώθηκε με νόμο τον 4014 το 2011 αλλά το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν το ε, αναμενόμενο. Αντί να η νομοθεσία να αποσαφηνίσει, περιέπλεξε ακόμη περισσότερο το ζήτημα. Καταρχήν, ο εθνικός νομοθέτης δεν αναγνωρίζει ότι η διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφος 3 και 4 είναι ειδική και διακριτή σε σχέση με αυτή δύο άλλων οδηγιών της, ε, οδηγίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οδηγίας για την ε, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αλλά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πάγια νομολογία του έχει κρίνει ότι η διαδικασία που θεσπίζει το ωσάνο άρθρο είναι διακριτή τόσο από τη διαδικασία της οδηγίας, όσο, ε, της, ε, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και από εκείνη της οδηγίας της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης. Με το άρθρο 10 του νόμου 4014 του ελληνικού νόμου δηλαδή επιβάλλεται η υποβολή ειδική οικολογικής αξιολόγησης στην αδειοδοτούσα αρχή για τα σχέδια των κατηγοριών α και β ως προς τον τύπο της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης προβλέπεται ότι οι έργα της, ε, μιας κατηγορίας μπορεί να αποτελούν ε, αυτή η εκτίμηση τμήμα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενώ σε άλλα έργα ε, υποβάλλεται αυτοτελώς. Οι, οι παραπάνω <clears throat> ρυθμίσεις δεν ενσωμάτωσαν σωστά τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 9243 όπως αυτές ερμηνεύτηκαν από το ε, Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, από αυτά φαίνεται κατά την άποψη μας των νομικών κάποιων Ελλήνων νομικών ότι από αυτά αποτελούν παραβίαση των οσάνου διατάξεων της εν λόγω οδηγίας. Προβληματική είναι επίσης και η ρύθμιση του άρθρου 11 του νόμου 4014 ε, που οι προβλέψεις του είναι αντίθετες με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, δηλαδή της οδηγίας 92-43. Γιατί το δικαστήριο το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ε, οποιοδήποτε έργο ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τις διαστάσεις του πρέπει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Ε, τέλος και κλείνω λόγω χρόνου είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχει θεσπιστεί μια ε, ανεξάρτητη περιβαλλοντική αρχή ανεξάρτητη από την αδειοδοτούσα αρχή η οποία θα αξιολογεί τη δέουσα εκτίμηση. Σας ευχαριστώ και θα μου δώσετε την ευκαιρία να επανέλθω αργότερα. Θα καταθέσουμε έγγραφα τα οποία περιέχουν πολλά περισσότερα από αυτά που κατόρθωσα να πω σε πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο σας. Ο κύριος Αδαμόπουλος. Για πέντε λεπτά και αυτός. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, αφήστε μου, επιτρέψτε μου να σχολιάσω. Το θέμα για το λόγο για τον οποίο οι σκουριές έγιναν γνωστές και εκτός του ελληνικού κράτους είναι διότι δεν είναι μόνο ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Οι σκουριές θυμίζουν ότι ο αγώνας για ένα πιο πράσινο και καθαρό πλανήτη είναι ένας αγώνας για την ανθρωπότητα, μια, ένας δίκαιος αγώνας. Το περιβάλλον είναι χώρος παγκόσμιας διακυβέρνησης, όπου κανένα κράτος, διακυβέρνηση ή άτομο δεν μπορεί να παρέμβει μόνο του και όπου κανείς δεν παραμένει ανεπηρέαστος. Το περιβάλλον μας δεσμεύει με άνευ προηγουμένου τρόπο διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης. Οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Βραζιλία, την Αυστραλία, η αύξηση του επίπεδου της ε, θάλασσας, η υπεραλίευση, η εξόριξη, η εναπόθεση τοξικών ουσιών επηρεάζουν όλους μας. Δεν, πρέπει να επιτρέψουμε να κληρονομήσουν κάτι τέτοιο οι επόμενες γενιές. Οι σκουριές δεν είναι το ανάθεμα της Χαλκιδικής, είναι η είναι το γεγονό ότι δόθηκε προτεραιότητα στην ανάπτυξη τη Ελλάδος ει βάρο του περιβάλλοντος και της ζωής. Οι σκουδιέ είναι, αφορά κάτι ακόμα πιο δυσάρεστο, μια δυσάρεστη αλήθεια, την αλήθεια του κρατικού εγωισμού, της έλλειψης διαφάνειας, των ε, εκπιπτών των ε, θεσμών της, ε, του κράτους, την, ε, τον ανελαίητο τρόπο με τον οποίο οι κρατικές ελίτ πουλούν τον δημόσιο πλούτο, που θέτουν σε κίνδυνο τις ελευθερίες και την υγεία του καθενός, ρηπαίνοντας και που αποτελούν έναν βασικό κίνδυνο της, των οικοντόπων, της πανίδας, της χλωρίδας και της ανθρώπινης ζωής. Ο αντίκτυπος των εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε κάτι που είναι μια περιοχή που ήδη υφίσταται κίνδυνο σεισμικούς θα, έχει, θα οδηγήσει απώλεια ε, 130.000 στρεμάτων δάσους και ε, ο όγκος της σκόνης θα είναι, που θα παραχθεί θα είναι τεράστιος. 480.000 κυβικά μέτρα νερού θα αντλούνται ανά ώρα με φοβερές συνέπειες στην, στα υπόγεια ύδατα που θα μειωθούν κατά 600 μέτρα τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα θα ρηπανθούν από θιούχα ε, οξέα και τοξικά ε, μέταλλα που, θα, που είναι δηλητηριώδη ακόμα και σε μικρές ποσότητες. Πώς μπορούμε να μην αμφισβητήσουμε τον αντίκτυπο της παρέμβασης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. Πώς μπορούμε να αρνηθούμε έμεσα ή άμεσα στο δικαίωμα την, ε, στις τοπικές κοινότητες της και την ανθρωπότητα συνολικό το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τις κυβερνήσεις τους. Μετά την ακρόση αυτή της αναφοράς, της 9 πριν από τρία χρόνια, ο Δήμος του Αριστοτέλη έστειλε τη γνωμοδότησή του, όπου υπογράμμισε ότι η εξορρυκτική δραστηριότητα προσβάλλει την αρχή της βιωσιμότητας και δεν διασφαλίζει με δίκαιο και ξεκάθαρο τρόπο το περιβάλλον, την, ε, τις κοινότητες και την οικονομία. Δυστυχώς, δεν, λαβ, δεν η, η, απόφαση αυτή δεν λήφθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υγείας της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής αυτής, η παρουσία μου εδώ σήμερα είναι, αποτελεί έκκληση για την καταγγελία της περιβαλλοντικής καταστροφής της Χαλκιδικής. Έκκληση να κρατηθεί αυτή η αναφορά ανοιχτή, διότι η Οδηγία 9243 και 147 του 2009 παραβιάζονται και ζητώ να ζητηθεί από την, από την ελληνική κυβέρνηση γνωμοδότηση για την εξέλιξη αυτή και, για, να, και να δημιουργηθεί μια νέα μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου. Κάνω έκκληση να επισκεφθείτε την περιοχή με αντιπροσωπεία σας για να δείτε και την περιβαλλοντική καταστροφή αλλά και την κοινωνική διαίρεση που έχει δημιουργήσει το έργο αυτό. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να σας ε, να τελειώσω με τα λόγια η Ερυσός, η ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Γαλλική Λιμπερασιόν το 2013. Την ιστορία αυτών των ανθρώπων επέλεξαν μια στάση περήφανη και αποφασισμένη. Θα πρέπει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για όλες τις γυναίκες και για όλους τους άνδρες που φιλοδοξούν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη βαρβαρότητα των αγορών. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you very much indeed, Madam Chair. Thank you, Miss. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δαμόπουλε. Θα ακούσουμε τώρα την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. κύριος Γιάννης Κουνινιώτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με πολύ ενδιαφέρον ακούσαμε τα σχόλια και τα επιχειρήματα των αναφερόντων και τους ευχαριστούμε. Σημείωσα επίσης ότι θα μας δώσετε και περαιτέρω γραπτά σχόλια. Θα τα μελετήσουμε με προσοχή. Θα ήθελα να πω ότι σμεριζόμαστε τις ανησυχίες των αναφερόντων. Πράγματι, ακριβώς η ίδια η φύση αυτού του σχεδίου, αυτού του έργου θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει επαρκής εξέταση και εκτίμηση, δέουσα εκτίμηση της λειτουργίας αυτού του έργου Υπάρχουν λοιπόν δυνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ε, και ίσως και γι' αυτό έχουν υπάρξει τόσες ε, διαδικασίες ενώπιον ε, των ελληνικών δικαστήριων για ακύρωση αυτού του έργου και υπάρχουν κάποιες ακόμη που δεν έχουν εκδικαστεί, δεν γνωρίζουμε δηλαδή πότε θα τιμιγορήσει το δικαστήριο για ορισμένες προσφυγές. Ήδη από το 2013 το Συμβούλιο Επικρατεία σε μια πρώτη του απόφαση είχε αποφασίσει πως η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην οδηγία για τα οικοσυστήματα, του σκοτόπους και για την περιοχή περιβαλλοντική εκτίμηση επιπτώσεων, τη διατάξη αυτών των δύο οδηγιών είναι, γίνονται σεβαστέ, άρα έχει υπάρξει επαρκής μελέτη, δέουσα μελέτη. Βέβαια, στο πλαίσιο των δημόσιων διαβουλεύσεων ακούστηκαν πολλέ και διαφορετικέ απόψει. Ε, κάποιε μελέτε προβάλλουν κάποια προβλήματα, κάποιε θεωρούν ότι δεν υπάρχει αντίκτυπο. Όπω καταλαβαίνετε πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο έργο και υπάρχουν και αποκλίνουσε απόψει ενίοτε. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το Συμβούλιο Επικρατείας είχε ε, μελετήσει, είχε εξετάσει μια πρώτη μελέτη αντικτύπου, όπου οι ελληνικές αρχές ε, ε, έλεγαν ότι μόνο 0,04% θα ήταν ο αντίκτυπος και όχι σε προτεραιότητας οικοσυστήματα. Οπότε είχαν θεωρήσει πως ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και σε σχέση με το δίκτυο Natura 2000 θα είναι απειροελάχιστη ο αντίκτυπο. Φυσικά αυτό είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία. Υπήρχε και μια πιο πρόσφατη απόφαση, πολύ πιο πρόσφατη από το ίδιο όργανο την προηγούμενη εβδομάδα που ακυρώνει υπουργική απόφαση και καταλήγει στο ότι το εν λόγω έργο μπορεί να προχωρήσει. Και όπως σας είπα υπάρχουν και άλλες υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί και περιμένουμε να ακούσουμε και τι θα αποφασίσει και το ανώτατο δικαστήριο. Εμείς από πλευράς Κομισιόν θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Είναι ένα σημαντικό έργο όπως είπα και πράγματι μπορεί να έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο αν δεν εφαρμοστεί με τον ε, δέοντα τρόπο. Παράλληλα όμως θα πρέπει να σεβαστούμε και την ετοιμιγορία ε, των δικαστηρίων ε, και στην προκειμένη περίπτωση του ανώτατου δικαστικού φορέα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Εδώ τώρα μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση, να ακούσουμε τους βουλευτές που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο. Η κυρία Ουκεν είναι η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ εκπλήσωμαι, πραγματικά. Είναι σαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείχνει πολύ μεγάλη απροθυμία ε, και ε, ξέρουμε ε, ότι αν αρχίσουμε να μελετάμε σε βάθος ε, τα θέματα των εξορίξεων, ιδίω ό,τι αφορά την εξόριξη χρυσού, θα βρούμε πολλά και διάφορα. Εδώ και χρόνο το συζητούμε το θέμα αυτό. Και από ό,τι φαίνεται όλα έγιναν λάθος, όλα πήγαν στραβά. Αλλά τι κάνουμε τελικά. Αντιδρούμε όταν πια δεν υπάρχει τίποτα να διορθωθεί. Και νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πολύ περισσότερο για τρεις λόγους τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε να γίνει σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία και το περιβαλλοντικό δίκαιο, που πραγματικά το περιβάλλον πάντοτε ε, δέχεται απειλέ. Πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική η Ένωση. Επίσης ε, δεν έχει γίνει σεβαστή σύμβαση του άρχους ε, και οι αναφέροντες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα έχει γίνει σεβαστή κατά την άποψή σας λοιπόν η σύμβαση αυτή. Και κάτι άλλο. Θεωρείτε, στην Κομισιόν στρέφομαι, θεωρείτε ικανοποιητικό αυτό να λέτε ότι έγινε μια μελέτη αντικτύπου και ναι, ε, μάλλον θα είναι πολύ περιορισμένος ο αντίκτυπος, αν μπορεί να είμαστε και σίγουροι κτλ. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε, αλλά παρακολουθούμε την κατάσταση. Μα είναι δυνατόν. Με τέτοια στρατηγική μπορεί να δημιουργηθεί σεβασμός γύρω από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εμείς γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα ε, τα χρυσορυχεία και στη Βουλγαρία έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μείνει ανίσχυροι τελικά αν απεμπολίσουμε όλα τα εργαλεία και ε, όπλα που έχουμε για να απαντήσουμε ε, στις πολύ θεμητές ανησυχίες των πολιτών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, πραγματικά πιστεύετε ότι έχει γίνει σεβαστή εδώ ευρωπαϊκή νομοθεσία? Γιατί αυτή είναι η οποία υπερτερεί η νομοθεσία και ο σεβασμός της. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Σε ευχαριστώ, Μαργκρέτε. Κύριος ε, Βίντσε. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η εξόριξη του χρυσού, τα ορυχεία χρυσού, προκαλούν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αν δούμε τι γίνεται στη χώρα μου, τι συνθήκες επικρατούν στη χώρα μου. Το 2000 είχαμε μια καταστροφή, περιβαλλοντική καταστροφή. Και επηρέασε και τη Ρουμανία και την Ουγγαρία αυτή η καταστροφή. Σαν αποτέλεσμα, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα. Και αυτό οδήγησε σε σχέδια εξέτασης των συνεπειών ε, της εξορίξεως του χρυσού και των χρυσορυχείων διότι οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στα χρυσορυχεία ε, ελοχεύουν, ε, έχουν πολλούς ε, κινδύνους στο περιβάλλον, κυρίως μέσω της παραγωγής ρηπαντών. Και αλλάζει και το τοπίο, προφανώς. Οι εικόνες λοιπόν που είδαμε μας το έδειξαν τέλεια την αλλαγή του τοπίου. και συμπεριλαμβανόταν και τοποθεσίες ε, Natura 2000. Έχουμε και την άλλη όψη του νομίσματος βεβαίως. Είναι θεμητό οι χώρες να θέλουν να εκμεταλλευτούν τα χρυσορυχεία. Αν δούμε όμως τα οικονομικά ωφέλη από τη μια και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και να δούμε τη σχέση μεταξύ τους και πώς επηρεάζονται και τα τοπία και οι άνθρωποι και η ζωή των ανθρώπων, βλέπουμε ότι αυτός ο αντίκτυπος αρνητικός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Προφανώς πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας επί του περιορισμού των κινδύνων. Αν δούμε τώρα τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν, πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να δράσει στεναρά και να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα όσον αφορά το περιβάλλον. Συνεπώς, συμφωνούμε ότι αυτή η αναφορά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Επόμενος, ο κύριος Αρβανίτης παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Όταν είχε έρθει η κυρία Σκακέλερ στην περιοχή, είχε μείνει άναυδη όσοι έχουν έρθει στην περιοχή έχουν μείνει άναυδοι. Έχω πάει, η εργασία μου πριν ήταν δημοσιογράφος, έχω καλύψει το θέμα αυτό. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή που αφορά στο περιβάλλον, στους ανθρώπους, στον πολιτισμό, στην κληρονομιά, παντού. Πόσο αξίζει η ζωή. Πόσους κόκκους χρυσού αξίζει. Και να το δούμε και ανάποδα, πρέπει να σας πω ότι η, η καταστροφή στον, στον υδροφόρο ορίζοντα, η καταστροφή στο θαλάσσιο περιβάλλον, η καταστροφή στα χωριά δεν μπορεί να ισοσκελιστούν με 600 ή και με 1000 θέσεις εργασίας. Υπάρχει ένα τραγούδι στην Ελλάδα που λέει ότι για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Θεωρώ ότι, για να μην σας κουράσω, συμφωνώντας με τους συναδέλφους μου και με τον συνάδελφο από το Λαϊκό Κόμμα και πήρα πολύ αισιοδοξία με την οπτική που βλέπουν οι συνάδελφοι το θέμα μας. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα που δεν αφισβητεί κανείς, έτσι κι αλλιώς. Έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, των πολιτών. Υπάρχουν κυβερνητικέ ευθύνε για την επένδυση αλλά και για τις καθυστερήσεις, για την προηγούμενη κυβέρνηση λέω, αλλά και για τις καθυστερήσεις και τώρα είμαστε σε ένα νέο περιβάλλον όπου κλείνεται το μάτι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να στείλουμε παρατηρητέ, να, να, να, έρθουν οι άνθρωποι από την να πάει το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντο, να μείνει το θέμα ανοιχτό, να πάνε παρατηρητέ δικοί μα εκεί, να το δείτε. Και να δούμε αν αυτό έχει σχέση με αυτό που λέμε ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον. Στην κρίση που ζούμε σήμερα, στην περιβαλλοντολογική. Εδώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγκεκριμένη Επιτροπή ε, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί θέλω να σημειώσω και ένα τελευταίο. Ό,τι γίνει, Πρόεδρε, στην Χαλκιδική στις Κουριές θα ξεκινήσει αύριο δίπλα στη Θράκη και πιο πάνω στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε χθες. Σας ευχαριστώ. Thank you. Next to speak is... Κύριος Νικολάου Λαβάνος, επόμενος ομιλητής. Εξόρυξης χρυσού στις Κουριές, γενικότερα στη Χαλκιδική, από το μονοπόλιο της Ελληνικός Χρυσός, δεν είναι πρώτη φορά που απασχολεί την Επιτροπή Αναφορών. Μετά την αποδοχή της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων χρυσού από την Ελληνικό Χρυσός από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στα πλαίσια της πολιτικής στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτό που κάνει είναι να επιχειρεί να κλείσει τα ανοιχτά ζητήματα που έχει δημιουργήσει η λαϊκή παρέμβαση εκεί. Οι κινητοποιήσει των κατοίκων, των σωματείων, των εργατικών κέντρων της περιοχής, οι ερωτήσεις που έχουν καταθέσει στο, στην Ελληνική Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που κατά τα άλλα, κατά τα άλλα εμφανίζεται σαν υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος, με τη στάση που παίρνει επί της ουσίας αυτό που κάνει είναι να συνενεί σε ένα έγκλημα με τεράστιες προεκτάσεις στο φυσικό περιβάλλον όπως αποκαλύπτουν και οι ομιλίες των ε, αναφερόντων και τα υποστηρικτικά ε, έγγραφα που έχουν καταθέσει στην υγεία των κατοίκων της περιοχής αφού το σχεδιασμένο έργο σύμφωνα με εκτιμήσεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων άλλων επιστημονικών φορέων μπορεί να επιβάλλει μία αναστρέψιμες αλλαγές σε όλους αυτούς τους τομείς Διαψεύδονται οι διαβεβαιώσει τη Ελληνικό Χρυσό ότι στηρίζει την τοπική κοινωνία, όταν και στην πλειοψηφία του οι εργαζόμενοι τη εργάζονται σε επικίνδυνε συνθήκε, με χαμηλού μισθού, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα. Βεβαίω, σε εναρμόνιση βέβαια με τι κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για ελαστικέ σχέσει απασχόληση και τι αναδιαρθρώσει των εργασιακών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Αυτά εφαρμόζει και η επιχείρηση η παραπομπή του ζητήματο για διευθέτηση στο συμβούλιο τη επικρατεία μπήκαν και κάποια στοιχεία στη συζήτηση αποκρύπτει ένα βασικό θέμα ότι το δικαστικό σύστημα είναι ταξικό ε, αποφασίζει υπέρ συνήθω των μονοπωλιακών ομήλων και δικαιώνει τι απαιτήσει του. Ιδιαίτερα όταν κρίνονται τεράστια συμφέροντα, σύμφωνα με ασφαλείς εκτιμήσει στο υπέδαφο τη περιοχή, ε, βρίσκονται 160 τόνοι χρυσού, όταν τα αποθεματικά που έχει η Τράπεζα τη Ελλάδο είναι 149 τόνοι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αποφάσεις που παίρνονται στην πράξη νομιμοποίησαν και εκβιασμού τη επιχείρηση, ότι αν δεν γινόταν αυτό θα απολύσει εργαζομένους, ότι η μη παραχώρηση του έργου στις Κουριές θα οδηγήσει στο κλείσιμο δύο ακόμη μονάδων που διατηρεί σε άλλες θέσεις στην ίδια περιοχή. Συνεχώς έρχονται στο προσκήνιο νέες επιπτώσεις που έχει συνολικά η εξόριξη χρυσού σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Επί παραδείγματι, στις μεγάλες νεροποντές του περασμένου φθινοπόρου η ροή των ρεμάτων τη περιοχή συμπαρέσυρε επικίνδυνα απόβλητα από του χώρου απόθεση τη μονάδα κυρίω τη Ολυμπιάδα, με κίνδυνο μεταφορά τοξικών υλικών και μόλυνση των υδάτων και των επιφανειακών. Τα έργα τη Ελληνικού Χρυσό, με τι προβλέψει που έχουν για χώρο υγειονομική ταφή επιβλαβών ε, επικίνδυνων αποβλήτων, για επιφανειακή απόθεση ξηρού υλικού σε κήτε ρεμάτων, για δημιουργία φραγμάτων απόθεση πάνω σε ενεργά σεισμογόνα ρήγματα, είναι ορολογιακή βόμβα αυξάνεται συνεχώ ο κίνδυνο ενό τεχνολογικού ατυχήματο. Θα επηρεάσει αυτό σοβαρά την υγεία των κατοίκων, οι οποίοι ακόμα και σήμερα και με τα σημερινά δεδομένα αντιμετωπίζουν τι συνέπειε τη εξορρυκτική δραστηριότητα. Δονήσει, τρανταγμοί, επιβάρυνση τη γεωργία, τη κτηνοτροφία τη περιοχή από τα απόβλητα. Το ΚΚΕ λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τι ανισχύε των φορέων τη περιοχή. Έγκαιρα διοργανώσαμε ημερίδα για αυτά τα ζητήματα. Κατά την άποψή μα, η επένδυση στι κουριέ για του λόγου που έχουμε εκθέσει, είναι αντιλαϊκή και είναι και καταστροφική για το περιβάλλον. Θα μπορούσε να είναι αλλιώ. Εμεί λέμε βεβαίω. Βεβαίω θα μπορούσε να είναι. Στο πλαίσιο τη κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, όπου δεν θα καθορίζει την εξόριξη το κριτήριο του επιχειρηματικού κέρδου, το οποίο δεν υπολογίζει ούτε το μισθολογικό, ούτε το περιβαλλοντικό κόστο, δεν υλοποιεί τι αναγκαίε τεχνολογίε προστασία και προφύλαξη, αλλά το κριτήριο τη ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Πρόκειται κατά την άποψή μα για σύντημα σφοδρή αντιπαράθεση μαζικών φορέων με την κυβέρνηση και το μονοπόλιο της Ελληνικός Χρυσός, πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά, να διερευνηθεί το ζήτημα και με τα νέα στοιχεία που καταθέτουμε και να αναγνωριστούν οι δίκαιες ανησυχίε των κατοίκων και των μαζικών φορέων τη περιοχής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νικολάου. Ο κ. Άγγιος Σαλίβα. Να ευχαριστήσω και εγώ καταρχά του αναφέροντες που ήρθαν να υποστηρίξουν την αναφορά του. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους όταν λένε ότι συζητούμε θέματα περιβαλλοντικής ε, βλάβης, ψήλωση των δασών, όπως ακριβώς αυτά που βλέπουμε στις σκουριές. Και ότι αυτό δεν είναι ένα ελληνικό πρόβλημα μόνο, αλλά ένα παγκόσμιο και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Για το λόγο αυτό πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση, στέλνοντας επιστολή στην ελληνική αντιπροσωπεία, ζητώντας περι, λεπτομέρειες. Να, πρέπει επίσης να στείλουμε την αναφορά αυτή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για περαιτέρω ενημέρωση και να την κρατήσουμε ανοιχτή, ασκώντας πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση. Να πω και εγώ δύο λόγια Η Επιτροπή στηρίζεται σε δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ελλάδα και το προσωπικό μας παρακολουθεί αυτό το scoreboard του 19 για να αντιμετωπίσει τις διοικητικές υποθέσεις στην Ελλάδα σε πρώτο βαθμό σε δεύτερο, ε, ε, 700 σε τρίτο επίπεδο χίλιες υποθέσεις κατά μέσο όρο 2.200 ημέρες απαιτεί μία δίκη στην Ελλάδα, 6 χρόνια δηλαδή. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο να περιμένουμε 6 χρόνια γι' αυτό. Το θέμα πρέπει να λυθεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και με βάση και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι η Επιτροπή και η Ένωση συνολικά δεν μπορούν να αποστούν από το πρόβλημα αυτό. Συμπέρασμα. Δύο λεπτά για τους αναφέροντος. Ο κ. Παναγιωτόπουλος δύο λεπτά, ο κ. Αδαμόπουλος δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ε, γνωρίζουμε ότι τέτοια θέματα αντιμετωπίζονται από τα εθνικά δικαστήρια καταρχήν. Η αναφορά μας στοχεύει στο ότι η εθνική νομοθεσία δεν ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία στα συγκεκριμένα θέματα. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο δηλαδή, αποδέχεται την εθνική νομοθεσία και όχι την ευρωπαϊκή. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πάρα πολλές υποθέσεις που αφορούν τέτοιου είδους δραστηριότητες αργεί πάρα πολύ να βγάλει αποφάσεις ή να εκδικάσει τις αποφάσεις, τις ε, υποθέσεις αυτές. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που καταθέσαμε αυτή την αναφορά στην Επιτροπή σας. Γνωρίζουμε τις αρμοδιότητες και των εθνικών δικαστηρίων και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και των επιτροπών του, της Ευρωβουλής. Ε, θα, κάνω και, θα κάνω και εγώ εκπροσωπώντας όλους τους υπογράφοντες την ε, αναφορά αυτή να παραμείνει και να εξεταστεί η υπόθεση αυτή στην ε, Επιτροπή σας και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και καλό θα ήταν μια ομάδα, μια αντιπροσωπεία να επισκεφθεί την περιοχή, να δει πώς είναι, να μιλήσει με ανθρώπους, να μιλήσει με επιστήμονες που για μια δεκαπενταετία ή για μια εικοσαετία ασχολούνται με το πρόβλημα των μεταλλίων της Χαλκιδικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας Επιστρέφω και 10 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ και πάλι. Thank you. Three seconds. Τρία δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αδαμόπουλος, Σωτήριος Αδαμόπουλος, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν θα χρησιμοποιήσω τα δύο λεπτά, απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την υποστήριξη που δώσατε στην αναφορά μας σήμερα. Χαίρο διότι βλέπω μια διακομματική συμφωνία από ό,τι καταλαβαίνω για το θέμα. Θέλω να κλείσω τη σημερινή μου τοποθέτηση παραθέτοντας την έκθεση του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που περιέγραψε τον αντίκτυπο της εξωεκτικής δραστηριότητα στην περιοχή ως σημαντική, αναπόδραστη και καταστροφική. Ευχαριστώ. Κλείνουμε νομίζω το θέμα αυτό. Υπάρχει ομοφωνία. Δεν μας αρέσει το γεγονός ότι η Επιτροπή κρύβεται πίσω από την αναζήτηση τοπικών λύσεων. Πρέπει να δουλέψετε περισσότερο. Η πρότασή μας είναι δεδομένου του μεγέθους του έργου και της πιθανότητας περιβαλλοντικού αντικτύπου, ζητάμε από την Επιτροπή να επανεξετάσει το θέμα μαζί με τους αναφέροντες, ιδίως να επανέλθει Ενημερώνοντα μα ενημερώνοντάς μας για το κατά πόσον ή ε, το έργο συμμορφώνεται με την οδηγία και την στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. Κατά την άποψή μου, ε, αν ε, ε, νομίζω ότι οι ομάδες δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα συναφή έγγραφα. Τουλάχιστον από όσο θυμάμαι δεν μας είχαν δοθεί τα έγγραφα και αυτό είναι παραβίαση της σύμβασης με, το, με την Κομισιόν. Του δύο και για τη μελέτη περιβαλλοντικού του 2001 και με τη σύμβαση του Όρχους. Να το σημειώσει αυτό η Επιτροπή. Ομά, ομόφωνη είναι η απόφαση της Επιτροπής. Ήρθε η πρόεδρος μας και της δίνω το λόγο για να συνεχίσει να προεδρεύει στη συνάντηση. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Είχε κακό καιρία στην Ισπανία. Συνεχίζουμε. Σημείο 6. Θα μιλώ Ισπανικά. Αναφορά 668-2018 από Βούλγαρο πολίτη για την παραβίαση του πιθανή παραβίαση του κανονισμού 1698 του 2005 της Ένωσης και της Οδηγίας 2009-28 από πλευράς του βουλγαρικού κράτους. Δεν είναι παρόν νομίζω ο αναφέρον, άρα δίδω το λόγο στην Επιτροπή. Στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, ο κύριος Πιέδρο Αέκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τη δυνατότητα να απαντήσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αναφορά το ιστορικό. Εν τη απουσία του αναφέροντος ισχυρίζεται ότι η Βουλγαρία δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου για να μην υποστηρίζει ανανεώσιμες εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας και θεσπίζοντας νέες τιμές στα πλαίσια των νέων προγραμμάτων να πω ότι υποστηρίζει πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρχή που περιγράφει ο αναφέρον. Δηλαδή τα κράτη-μέλη όταν σχεδιάζουν υποστηριχτικά σχέδια θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι είναι σταθερά και παρέχουν μέγιστη προβλεψιμότητα και ορατότητα για τους επενδυτές ούτως ώστε το κόστος της ενεργειακής μετάβασης να είναι το χαμηλότερο δυνατό. Είναι αρχή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει επανειλημμένα και είναι γεγονό ότι η αναδιατύπωση της οδηγίας περανεωσίμων που υιοθετήθηκε το 2018 έχει ένα νέο άρθρο που απαιτεί από τα κράτη-μέλη, από, μάλλον αποτρέπει τα κράτη-μέλη από τροποποίηση των υποστηρικτικών του ε, συστημάτων που αναδρομικά θα επηρέαζε αρνητικά ε, υφιστάμενα δρομολογηθέντα προγράμματα. Το 2018 λήφθη η απόφαση αντιτύπωση τη οδηγία για τα ανανεώσιμα ή τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Τώρα, για την αναφορά τη συγκεκριμένη. Πρέπει να αναλυθεί στα πλαίσια τη ισχύουσα οδηγία για ανανεώσιμε και τη προηγούμενη του 2008. Σε αυτή την οδηγία είναι σημαντικό να θυμηθούμε δύο πράγματα. Τα κράτη-μέλη υπέχουν νομική υποχρέωση μέχρι το 2020 να έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανανεωσίμων στο ενεργειακό μείγμα. Στη Βουλγαρία έχουμε 16%. Άλλη υποχρέωση. Μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν που έχουν σχεδιαστεί ούτω ώστε να εξασφαλίζουν ότι ενώ καθοδόν προς το 2020 θα ακολουθείται μια συγκεκριμένη τροχιά και πορεία. Δύο πράγματα συμπεραίνουμε από αυτά. τα κράτη-μέλη δεν έχουν αυτά καθεαυτά υποχρέωση να έχουν υποστηρικτικά μέτρα για την ε, ανανεώσιμη ψυχή ενέργεια. Είναι ένα από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν τι ανανεώσιμε ψυχέ ενέργεια. Δεν έχουν υποχρέωση να έχουν συγκεκριμένα σχήματα και συστήματα. Η Βουλγαρία μετά είναι πάνω από την προκαθοριστή απορία της οδηγίας και το 2017 είχε ξεπεράσει το επίπεδο που απαιτείται για το 2020. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεραίνει ότι Ουσιαστικά δεν υπάρχει παράβαση που απορρέπει την αλλαγή του συστήματος υποστήριξης, διότι δεν υπέχει χώρα πρώτης ε, νομική υποχρέωση να θεσπίσει ένα τέτοιο μηχανισμό και μετά τα μέτρα που πρέπει να σχεδιάζονται τόσο ώστε να εξασφαλίζουν ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό ανανεωσίμων είναι στο ενεργειακό μείγμα δεν εφαρμόζεται αυτό το πλαίσιο συγκεκριμένα εφόσον πληρεί τι προποθέσει και την αδεικτική πορεία προ το στόχο ήδη η Βουλγαρία. Τέλος, για τον ισχυρισμό, για παραβίαση ε, των προσδοκίμων, των ε, θεμητών προσδοκιών. Σύμφωνα με τον ομολογία, αυτή η αρχή δεν μπορεί ξεχωριστά να ερμηνεύεται, πρέπει να ερμηνεύεται σε συσχετισμό με συγκεκριμένη νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πέρα από τα εθνικά μέτρα. Δηλαδή, η υποχρέωση να υπάρχει ένα πλαίσιο υποστηρικτικό το δικαστήριο είπε ότι οι οικονομικοί φορείς δεν δικαιολογούνται να έχουν θεμητές προσδοκίες. Θα διατηρηθεί η φυστάμενη κατάσταση. Αν η κατάσταση μπορεί να αλλάχθεί από τις εθνικές αρμόδιες αρχές εν τη εκτελέση της διακριτικής τους δυνατότητας, κάτι που αναφέρεται στην ισχύουσα οδηγία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το λόγο έχουν οι εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ράντεφ μου ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αν με επιτρέπετε, θα ήθελα και εγώ εν συντομία να μιλήσω για αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τους αναφέροντες ότι αν ε, τερματιστούν οι επιδοτήσεις ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, η Βουλγαρία δεν θα τηρεί τις δεσμεύσεις που, και τις πόχες που υπέχει κατά το δίκαιο. Το 2009 και έκτοτε πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη ε, κάποιες διατάξεις, τα ΙΣΑΠΕ, μέχρι το 2020. Στόχος είναι να υπάρχει ε, ένα μερίδιο ε, του ενεργειακού μείγματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η οδηγία στηρίζει και την επιλογή κρατών μελών, την επιλογή των κρατών μελών, ε, έστω και ενός μέσου που θα επιτρέπει την συμμετοχή των ΑΠΕ στο μείγμα, το ενεργειακό. Για το 2017 η Eurostat έχει καταθέσει στοιχεία που δείχνουν ότι για το 2020 ξεπερνάμε ε, στην Βουλγαρία έναν δείκτη συγκεκριμένα. Και σε ό,τι αφορά το μερίδιο ΑΠΕ το 2017 για τη Βουλγαρία ήταν 18,7%. Πάνω από τον ενδεικτικό στόχο δηλαδή του 2015-2016 που ήταν 12%. Και ο στόχος για το 2020 είναι 16, που το ξεπερνάμε και αυτό επίσης. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το, τα κίνητρα για την ενεργική πολιτική και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, αυτά τα πρότυπα τηρούνται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αγορά ΑΠΕ. Η οδηγία του 9 δεν παραβιάζεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει στην απάντησή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2019. Έχουμε το άρθρο 3 παράγραφος 2 που θέτει τις προϋποθέσεις για το σχεδιασμό μέτρων όπως ε, μέτρα στήριξη και Και αυτή η προπόθεση είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εγγυώνται ότι το, μείγμα, το μερίδιο με την θα ισούται ή θα υπερβαίνει τον ενδεικτικό στόχο που αναφέρεται Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Βουλγαρία πληρεί ε, τι εν λόγω ε, προποθέσει. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι δικαιολογημένη η αναφορά και θα σαν να κλείσει. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Άουκεν. Κοιτάξτε, ε, λίγο παράλογα μας τα λέτε εδώ. Έγιναν εκλογές. Και ε, στο επίκεντρο της προεκλογικής καμπάνιας ήταν το κλίμα. Και τι ακούμε τώρα εδώ πέρα, ότι η Βουλγαρία λέει είχε αυτό το μετροπαθή στόχο το 18% σε σχέση με αυτό που τουλάχιστον φιλοδοξούμε να πετύχουμε. Και ο στόχος ποιος είναι τελικά. Να μην έχουμε αυτές τις ε, δυνατότητες και επιλογές. Και μας ενδιαφέρει το πώς επιδοτούνται οι άλλες πηγές ενέργειας που λέει και η Κομισιόν ότι για τον άνθρακα, για την πυρηνική ενέργεια. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα σε ό,τι τις Και εσεί ε, λέτε τώρα το αντάποδο. Να βρουν έναν άλλο τρόπο, λέτε. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε δηλαδή. Και λέτε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια ε, για τις επενδύσεις Γι' αυτό κάνουμε και νόμους, αγαπητέ συνάδελφοι. Γι' αυτό ακριβώς το σκόπο, για να υπάρχει ασφάλεια όταν επενδύουν ε, κάποιες βιομηχανίες, για να ξέρουν ότι δεν θα αλλάζουν στόχοι, δεν θα αλλάζουν τα συστήματα. Αυτός ο στόχος, λέει, είναι υψηλότερος. Είμαι χρόνια εδώ και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, αλλά πραγματικά εκπλήσωμαι που λέτε ότι έχουμε αυτό το 18% μέχρι το 2020 πριν το πετύχουμε, μα είμαστε ήδη στο 2020 τέλος πάντων και λέτε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι περισσότερο. Μα τελικά ο κίνδυνος να πάτε πίσω, να Μειώστε τις προσπάθειες και η Κομισιόν λέει σταματάμε φέτος γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Αντίθετα, η Κομισιόν θα έπρεπε να βοηθήσει τις χώρες να πετύχουν τους στόχους. Έχουμε και το πράσινο σύμφωνο. Εσείς λέτε θέλετε να κάνετε το αντίθετο όμως με βάση στρατηγική σας. Thank you. Uh, Danoka. Ευχαριστώ κυρία Ντανόκα. Και εγώ έχω εμπειρία από τη χώρα μου, τη Λετωνία. Πολύ μεγάλο το σκάνδαλο. Χρησιμοποιήθηκαν αυτού του είδους τα προγράμματα για μικρούς υδροελεκτρικούς σταθμούς και αυξήθηκε έτσι η τιμή της ενέργειας, μπορούσαν να αυξήσουν τη τιμή της ενέργειας χωρίς λόγους ουσιαστικούς και η κοινή γνώμη για την πράσινη πολιτική έγινε πολύ αρνητική. Αυτή η εφαρμογή εθνικών μέτρων εντάσσεται στην επικουρικότητα αλλά πρέπει να ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς εφαρμόζονται όλα αυτά. Απλή συμμόρφωση με εθνικούς στόχους δεν αρκεί. Αν αυτά τα μέτρα δεν ελέγχονται σωστά και δεν ευσταθούν. Εκεί πρέπει να εκφράζουμε ανησυχία. Και αυτό έκαναν οι αναφέροντες. Εμπιστεύομαι την ευαισθητοποίησή τους πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω το θέμα. Άρα να μην κλείσει η αναφορά. Ευχαριστώ. Και Σαλίβα. Η Βουλγαρία δεν παραβιάζει την οδηγία 28-2009. Η αλλαγή του στήματος υποστήριξη δημιουργεί ανησυχίε όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη προστασία των επενδύσεων που γίνονται από τους πολίτες τη Βουλγαρία. Γι' αυτό λαμβάνονται υπόψη επίσης το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κυρίως για την Πράσινη Συμφωνία, γι' αυτό πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Και η Επιτροπή Ήτρε θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά αυτή την αναφορά. Μας Ευχαριστώ. Έχοντας ακούσει την Επιτροπή δεν είναι εδώ, όπως είπαμε, αναφέρον και έχοντας ακούσει και τα μέλη του σώματος προτείνω να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά κανείς δεν πρότεινε κάτι πέραν ωστόσο από το να το κρατήσουμε ανοιχτό. Να ζητήσουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση και τη επιτροπή Ήτρε, εάν συμφωνείτε. Ωραία. Κλείνει το σημείο αυτό. Ε, Σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. 838 του 2018 του κ. Κλάους Σάμερ, Γερμανού πολίτη, για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών οχημάτων για, την, ε, για να μπορούν να πάρουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο. Είναι εδώ ο κ. Σάμερ. Καλώς ήλθατε. Σας δίνω το λόγο για 5 λεπτά για να παρουσιάσετε τις θέσεις σας. Κατόπιν θα ακούσουμε την Επιτροπή, κατόπιν του συναδέλφου και στο τέλο έχετε πάλι δύο λεπτά για να σχολιάσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα γερμανικά αν μου επιτρέπετε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Θα ήθελα να σας θυμίσω την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα μετά το τσουνάμι στην Ιαπωνία ε, που έπληξε το σύστημα ηλεκτροδότησης, ε, που ε, δημιούργησε μεγάλο blackout. Άρα το θέμα είναι ο ηλεκτρισμός εδώ και τότε η Ιαπωνία αναγκάστηκε να αντιδράσει και αποφάσισε στην αυτοκινητοβιομηχανία να αλλάξει το σύστημα της φόρτισης και να έχει πλέον αυτό το σύστημα της αμφίδρομης ροής ισχύω και σε περίπτωση που υπάρξει μια φυσική καταστροφή και υπάρχουν ε, κάποιοι σταθμοί φόρτιση σε ένα σπίτι να μπορούν ε, να τροφοδοτούν αυτοί οι σταθμοί και το δίκτυο. Εμεί στην Ευρώπη δεν έχουμε βέβαια πρόβλημα τσουνάμι. Ε, Έχουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό είναι θετικό ε, και αρκετές ε, τέτοιες ε, διαφορετικές πηγές. Αυτό είναι θετικό, όμως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οδηγούν και σε έλλειψη σταθερότητας στο δίκτυο. Έχω ερευνήσει και το κόστος που θα απαιτηθεί για τη σταθεροποίηση μόνο και μόνο για το δίκτυο ηλεκτροδότησης στη Γερμανία που είναι 1,2 δις και μόνο και έχουμε αυτό το νέο σύστημα που θέλω να σας παρουσιάσω, το V2G, το Vehicle to Grid, αυτή αφίδρομη ροή ισχύω από το όχημα προς το δίκτυο. Δηλαδή όχι μόνο να εφοδιάζεται το όχημα με ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά να μπορεί να βοηθήσει και την σταθεροποίηση του δικτύου ε, για την αποφυγή περίοδων εχμής ε, που μπορεί να οδηγήσουν σε blackout κτλ. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, εταιρείε, ε, όπως η Τσαντέμου για παράδειγμα, που έχουν βρει τέτοιες τεχνολογίες φόρτισης και τις χρησιμοποιούν όχι για την αποφυγή μόνο προβλήματος σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, αλλά και για τη σταθεροποίηση του δικτύου. Έχουμε λοιπόν το σύστημα φόρτισης, συνδυασμένο σύστημα φόρτισης, που ενώ την έχουμε στο μυαλό αυτή τη δυνατότητα, δεν έχουμε προχωρήσει, σε, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, τουλάχιστον ε, σε ε, πρακτική ε, ενίσχυση για τη δημιουργία τέτοιας τεχνολογίας. 10 εκατομμύρια τα επόμενα 10 χρόνια στη Γερμανία θα είναι ηλεκτροκίνητα. Αυτός είναι ο στόχος να κυκλοφορεί στο δρόμο. Και αυτό σημαίνει ε, ότι έχουμε αυτούς τους ε, Ασιάτες το 20% που μπορούν να βοηθήσουν με αυτούς τους νέους σταθμούς ε, φόρτς, με αυτήν την τεχνολογία, αλλά το 80% όχι. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή τα ηλεκτροκίνητα μη ασιατικά οχήματα στην Ευρώπη να συνεισφέρουν στη σταθεροποίηση του δικτύου. Και πραγματικά αυτό κατά τη δική μου άποψη είναι ένας παραλογισμός. Να μην κάνουμε σχετικές ρυθμίσεις για να έχουμε αυτά τα πρότυπα. Έχω ε, μιλήσει με τους εκπροσώπους τύπου μιας γαμικής αυτοκινητομηχανίας. Μου είπανε ναι, το μελετάμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια τυποποίηση, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας για να συμπεριλάβουμε αυτή την τεχνολογία στα σχέδιά μας. Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα πρέπει η πολιτική να παρέμβει, θα πρέπει η παραγωγή να τους επιβληθεί να λάβουν υπόψη τους αυτήν την τεχνολογία όταν θέλουν να προωθήσουν ε, την ηλεκτροκίνηση και να φέρουν πολλά ε, ηλεκτροκίνητα οχήματα ε, στους δρόμους. Γι' αυτό παρακαλώ να μην κλείσει αναφορά, να παραμείνει ανοιχτή και το θέμα αυτό να το δει και η Επιτροπή Ενέργειας με μια σχετική έκθεση, με μια γνωμοδότηση σε σχέση λοιπόν με το πρόγραμμα αυτό. Είναι και θέμα της ιδιωτική ε, του ιδιωτικού κλάδου. Στη Βρετανία υπάρχουν project για το V2G, για αυτή την αφίδρομη φόρτιση ή ροή ε, Και υπάρχει και μια νοπική δημοσίευση για τις αριθμιστικές προβλέψεις σε ό,τι αφορά την Βόρεια Ευρώπη. Το θέμα είναι να υπάρχουν αυτά τα δυνατό, αυτές οι δυνατότητες στο δίκτυο, δηλαδή να υπάρχει αυτή η λεγόμενη αμφίδρομη ροή ισχύω και θα πρέπει βέβαια η πολιτική να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα στη βιομηχανία να περιλάβουν τέτοιου είδους πρότυπα, να εξοπλίσουν ε, τα οχήματα και τους σταθμούς ε, με αυτή τη δυνατότητα. Και νομίζω ότι θα έπρεπε η Επιτροπή να επιληφθεί και παρακαλώ εκ νέου να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Σαμπίν Κρούμ έχει το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ τον αναφέροντα που επεξήγησε το θέμα. Η ηλεκτροδότηση των οδικών μεταφορών θα παίξει σημαντικότατο ρόλο για την μείωση των εκπομπών άνθρακα στι οδικέ μεταφορέ, Έχει τονιστεί αυτό και στην Πράσινη Συμφωνία. Επ' αυτής της βάσης αναμένεται ότι ο αριθμό ηλεκτροκινήτων οχημάτων στου δρόμου θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια και τι επόμενε δεκαετίες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα οχήματα πρέπει να ενταχθούν αποτελεσματικά στο σύστημα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό δημιουργεί και προβλήματα αλλά και ευκαιρίε. Αυτό που κουβεντιάζουμε σήμερα και που θέτει αναφέρον είναι ευκαιρίε που δημιουργούνται από τις, από τις υπηρεσίες που μπορούν να παράσχουν οι μπαταρίες των ηλεκτροκινήτων οχημάτων που σταθεροποιήσουν το ηλεκτρικό σύστημα, το ηλεκτρικό δίκτυο και τέτοια σταθεροποίηση θα γίνεται όλο και πιο σημαντική με μεγαλύτερο ποσοστό ανανεωσίμων που θα χρησιμοποιείται στο σύστημα. που θα χρησιμοποιούνται ανανεώσιμε για παραγωγή ηλεκτρική ε, ενέργεια. Ξέρουμε το θέμα αυτό για τη σύνδεση των οχημάτων στο δίκτυο, τι ρόλο που μπορούν να παράσχουν σχετικέ υπηρεσίε φόρτιση των οχημάτων αμφίδρομη και πώ μπορεί να γίνει αποτελεσματικότερη η χρήση αυτή. Το Δεκέμβριο του 2018 είχαμε του νέου κανόνε που θεσπίστηκαν από του συνομοθέτε. Καθορίστηκε πλαίσιο. Να υπάρχουν υπηρεσίε σύνδεση των οχημάτων με το δίκτυο. Να δημιουργηθεί μια αγορά όχι μόνο για να δημιουργηθούν οι τεχνικές δυνατότητες για αυτές τις υπηρεσίες, ναι, να, υπάρχουν, να υπάρχει παροχή των υπηρεσιών, αλλά υπάρχει και αγορά για χρήση των υπηρεσιών. Οι εμπορικές υπηρεσίες ήδη υπάρχουν, V2G, στην Ευρώπη. Έχουμε το NUVE στην Ολλανδία, που χρησιμοποιούν κυρίως τα ιαπωνικής τεχνολογίας οχήματα, όπως τα Nissan. Δεν μπορεί να εγκατασταθεί κάτι, κάποιο χαρακτηριστικό σε κάποιο όχημα, ηλεκτρικό όχημα και να μπορεί να παρεχει υπηρεσιε υπηρεσίες V2G το όχημα. Είναι πώς επικοινωνεί το ηλεκτρικό όχημα με το δίκτυο που γίνεται στο σημείο φόρτισης. Αυτό είναι το θέμα. Όπω είδαμε και στην παρουσίαση έχουμε δύο συστήματα ανταγωνιστικά. Το Σαντέμο, το Ιαπωνέζικο, που μπορεί να κάνει αμφιδρομή φόρτιση αρκετοί Ασιάτες κυρίως αυτο, ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα και συνδυασμένο σύστημα φόρτισης. Οι Ευρωπαίοι και οι Βορειοαμερικάνοι κατασκευαστές και πάντα υποστηρίζει κάθε σημείο φόρτιση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να προβλέπει στην νομοθεσία, στην οδηγία για αναλλακτικά καύσιμα, ότι δημόσια σημεία φόρτιση θα πρέπει να εξοπλισμένα κατάλληλα. Αν υπάρχει υποχρεωτική απέτηση τα ηλεκτρικά οχήματα να μπορούν να παράσχουν και υπηρεσίε από το όχημα προ το δίκτυο, θα σήμαινε de facto θα επιβάλλουμε υποχρέωση στα ηλεκτρικίνητα οχήματα να είναι συμβατά με το στάνταρ σαντέμου. Αλλά το βασικό στάνταρ είναι το CTS. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν Σαντέμου δεν θα μπορούν να φορτίσουν να εκφορτίσουν στα περισσότερα σημεία φόρτιση Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό. Στο CCS στο CTS δεν μπορούν να κάνουν αμφίδρομη φόρτιση σε αυτή τη φάση, αλλά θα αναπτυχθεί περαιτέρω το σύστημα και κάποιες ανακοινώσει είδαμε στον τύπο, κάποιε πληροφορίες, ότι αναμένεται ότι η οι υπηρεσίε οχήματος προς το δίκτυο θα μπορεί να γίνει μέσω του συνδυασμένου συστήματος φόρτισης μέχρι το 2025. Από νομοθετική πλευράς, να πω το εξή. Γίνεται αναθεώρηση των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τη σχετική οδηγία. Θα εξετάσουμε λοιπόν και το θέμα επικοινωνία τη μπαταρία του ηλεκτροκίνητου οχήματο με το δίκτυο ηλεκτροδότηση και το σημείο φόρτιση. Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιε ανάγκε υπάρχουν, που χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση για να έρθουν εμπόδια όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από το όχημα προ το δίκτυο. Ο συνάδελφο ξέρει περισσότερα και θα σα δώσει πληροφορίε. Κλείνοντα. Οι παροχέ υπηρεσιών από όχημα προς το δίκτυο θα είναι σημαντικές από το 2030 όταν η κριτική μάζα, η κρίσιμη μάζα ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα κυκλοφορεί. Πρέπει να δούμε όχι μόνο αυτές τις υπηρεσίες, αλλά και τις εφιούς φόρτισης, smart charging. Το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο με το που πριζώνεται δεν θα φορτίζει. Μπορεί να λαμβάνει υπόψη και άλλους παράγοντες ε, Άλλε περιστάσεις. Όταν βάζεις το αυτοκίνητο στην πρίζα, όταν επιστρέφεις, να μην υπερφορτίζουν όλοι όταν πριζώνουν το αυτοκίνητό του την ίδια ώρα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένα σύστημα ε, φιούς ε, φόρτισης του οχήματος. Ευχαριστώ. Has the floor. Τούλιους. Ο κ. Τούλιους έχει το λόγο για την Επιτροπή. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Μία παρατήρηση σημαντική νομίζω. Όταν μιλάμε για το smart charging και είναι σημαντικό η, ότι η εξυπνάδα του συστήματος είναι στο φορτιστή, όχι στο αυτοκίνητο. Όταν κοιτούμε λοιπόν την αναθεώρηση της οδηγίας θα πρέπει να δούμε τις διατάξεις για να εξασφαλίζουμε ότι οι φορτιστές είναι έξυπνοι και ότι μέσω των φορτιστών μπορούμε να διαχειριστούμε την φόρτιση και αποφόρτιση του οχήματος. Το βασικό λοιπόν εδώ είναι ο φωτιστής και όπως εξήγησε η Σαμπίνε, το σύστημα επικοινωνίας ε, με τη σύνδεση ε, με το αυτοκίνητο να υπογραμμίσω ξανά αυτό που είπε η Σαμπίν. Με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το CCS είναι το στάνταρτ που πρέπει να εγκατασταθεί και είναι ήδη εγκαταστημένο σε όλα τα σημεία φόρτωσης. Τον... Η υποχρεωτικότητα αυτού του συστήματος έγινε για... στην Ευρώπη έγινε για να υποχρεώσουμε όλους να έχουν μία βεβαιότητα ότι το σύστημα τους είναι απόλυτα διαλειτουργικό και θα χρησιμοποιείται στο μέλλον. Το CCS λοιπόν είναι νομοθετική απέτηση από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό το πρότυπο πρέπει να διατηρηθεί. Για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η διαλειτουργικότητα στην Ευρώπη. Βεβαίως είναι προφανές ότι το σύστημα που έχουμε θα πρέπει να μπορέσει να ενταχθεί και στο ευρύτερο πλαίσιο της αναθεώρησης των, και των συζητήσεων για τις εναλλακτικέ μορφές ενέργειας. Οι βουλευτές τώρα. Ο κύριος Βίντσε από το ΕΛΚ. Πρόεδρε, είναι πολύ τεχνικό το θέμα βέβαια και ήταν πολύ χρήσιμη η τελευταία εξήγηση από πλευράς Επιτροπής που την ευχαριστώ γιατί μας επιτρέπει να καταλάβουμε το ευρύτερο πλαίσιο. Υπάρχει ευρωπαϊκό πρότυπο για, τα για την σύνδεση των ηλεκτρικών οχημάτων. Απλώς πρέπει να δούμε σε μια προοπτική κάποιων ετών. Ίσως ο στόχος του 2030 να είναι πολύ αργά αν θέλουμε να ξανασκεφτούμε ολόκληρη την αρχιτεκτονική του ζητήματος διότι η Πράσινη Συμφωνία και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιταχύνουν τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων τα επόμενα έτη. Οι πολίτες θα παροτρύνονται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Προφανώς είναι σημαντικό η βιομηχανία να έχει μία βεβαιότητα για την πορεία που θα προχωρήσουμε και να επενδύουν σωστά στην έρευνα και καινοτομία. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει και διασύνδεση μεταξύ των διαφόρων παραγωγών στην Ένωση και των παραγωγών, των στην Ιαπωνία. Και το πλεονέκτημα της αυτοκινητοβιομηχανίας μας είναι ότι θα πρέπει να μπορούν να παράξουν αυτοκίνητα που θα έχουν πρόσβαση στην αγορά σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε ήδη μια συζήτηση για τους φορτιστές των έξυπνων κινητών, των smartphones. Είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και για τα αυτοκίνητα, για τους φορτιστές να μπει σε λειτουργία και ένας κανονισμός για τα αυτοκίνητα. Ας κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή την ε, αναφορά. Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Με την πράσινη συμφωνία ανοίγουμε πολλούς, ε, πολλές πόρτες και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι παροτρύνουμε έξυπνες προς έξυπνες λύσεις για όλο τον πληθυσμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο τον αναφέροντα για την παρουσίασή του και ευχαριστώ και την Επιτροπή. Έχουμε ένα νέο σύστημα, αλλά ένα νέο πρότυπο, αλλά πρέπει να έχουμε ανοιχτές διαδικασίες και προτείνω να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να την προωθήσουμε στην Ήτρα. Κύριε Άουκεν, συμφωνώ. Με εκπλήσει να προσθέσω ότι χρειάζεται να νομοθετούμε εμείς. Ο κλάδος θα πρέπει να δει πώς πρέπει να το κάνει. Μερικές φορές πραγματικά με εκπλήσει ότι εμείς ζητούμε να καινοτομήσουμε. Υπάρχουν χώρες που ακόμα νομίζουν ότι το περιβάλλον δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται ωστόσο στην αυτοκινητοβιομηχανία σε, σε κάποια κράτη-μέλη. Να το κρατήσουμε ανοιχτό και να το στείλουμε στις αρμόδιες επιτροπές στην Ήτρε ιδίω. και να δούμε μήπως χρειάζεται να νομοθετούμε περισσότερο εδώ. Ίσως. Αλλά αυτό με εκπλήσει. Ο αναφέρον, κύριε Σάμερ, Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο αυτό που είπε η Κομισιόν ε, να περιμένουμε ουσιαστικά 10 χρόνια και να έχουμε αυτά τα 8 εκατομμύρια οχήματα ε, στο δρόμο. Δεν είναι για μένα λογική αυτή η προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά ε, το πρότυπο Σαντέμο, δεν είπα ότι πρέπει να το αντιπαραθέσουμε με το ευρωπαϊκό. Απλά είπα ότι υπάρχει ήδη αυτό το πρότυπο και αυτό το πρότυπο Σαντέμο ε, λέτε ότι δεν λειτουργεί επί της αρχής. Όχι, λειτουργεί, γιατί υπάρχουν ε, οχήματα τα οποία ε, λειτουργούν με αυτό το σύστημα και μπορούν να φορτιστούν με αυτό. Και έχουμε μέχρι στιγμής 90% των ασιατικών οχημάτων που έχουν αυτό το σύστημα, αλλά δεν είναι πρόβλημα σταθμού φόρτισης και τεχνολογίας, αλλά τεχνολογίας του οχήματος. Δηλαδή, οι κατασκευαστές οχημάτων θα πρέπει, όπως και οι ε, ασιάτες, ε, αυτοκι... οι ασιατικές αυτοκινητοβιομηχανίες ε, να το κάνουν και εκ των προτέρων, γιατί ο εξοπλισμός εκ των υστέρων με αυτή τη διάταξη, με αυτό το εξάρτημα, θα είναι πάρα πολύ πιο δαπανηρό να έρθει όταν θα έχουμε ήδη 8 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη. Και κάτι ακόμη για την Κομισιόν, για αυτή την αφιδρομή φόρτιση, να περιληφθεί στο CCS. Αυτός είναι ο στόχος, αλλά αυτό μπορεί να χρειαστεί πέντε χρόνια να γίνει. Πρέπει λοιπόν τώρα να κάτσουν ε, οι αρμόδιοι με τις αυτοκινητομηχανίες ε, στο τραπέζι και να δούμε αν θα μπορούσαμε σε δύο-τρία χρόνια να έχουμε αυτό το πρότυπο. Να μην, παραλαμβάνω, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που θα έχουμε ήδη 8 εκατομμύρια χαζά, για να το πω έτσι, ηλεκτροκίνητα οχήματα τα οποία θα ε, κυκλοφορούν τότε στον δρόμο και προσπαθούμε εκ των υστέρων να τα εξοπλίσουμε. Πρέπει λοιπόν ε, να ε, γίνει μια ε, διατύπωση ενός προτύπου με αυτά ακριβώς τα οποία ζητώ και ελπίζω να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ τον αναφέροντα. Ακούσαμε λοιπόν και εσάς και την Κομισιόν και τους συναδέλφους μας, μέλη της, Αναφορών. Θα κρατήσουμε πράγματι ανοιχτή την αναφορά και θα ζητήσουμε και την γνώμη της Επιτροπής Ήτρε για να συνεχίσουμε να προχωρούμε σε αφορά την ανάπτυξη τροπο... Ε, νομοθεσίας για την προσαρμογή μας ε, στο ε, πράσινο σύμφωνο και για να προσαρμόσουμε τα οχήματα στις ανάγκες της εποχής. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο 854 του 2018 από Γερμανό πολίτη εξ ονόματος της ε, Γερμανικής Εταιρείας Φίλων των Σιδηροδρόμων για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τον φόρο εργασιών για τους διάφορους τρόπους μεταφορών τουριστικού χαρακτήρα. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον. Θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Στον κύριο Κουμπίτσα πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Ο αναφέρον ζητά δύο πράγματα. Είναι για το ΦΠΑ στις μεταφορές. Ζητά ειδικού συντελεστέ για ειδικού τρόπους μεταφοράς και δεύτερον εμέσως ζητά να αλλάξει ο, φόρος, ο χώρος φορολογίας. Σε ό,τι αφορά τους συντελεστέ. τα κράτη-μέλη μπορεί να έχουν είτε μειωμένο είτε τον κανονικό ΦΠΑ τώρα. Αυτή η ευελιξία υπάρχει αυτό που ζητά ο αναφέρον είναι δυνατόν, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουμε μηδενικό συντελεστή. Η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2018 πρότεινε νέου κανόνες για τους ε, συντελεστές αυτέ που δίνουν μεγαλύτερη ευελιξία και επιτρέπουν και μηδενικό συντελεστή. Θα μπορούσε σε μια τέτοια περίπτωση να υπάρχει μηδενικό συντελεστή για τις ε, σιωδρομικές μεταφορές, ε, μειωμένο για το λεωφορείο και κανονικό συντελεστή για τα, τις αερομεταφορές. Αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα και αφορά γενικότερα τους κανόνες για τους συντελέστέ. Ε, η κροτική Προεδρία θα συζητήσει το θέμα αυτό, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά θα πάρει χρόνο. Το δεύτερο ερώτημα είναι λίγο πιο σύνθετο. Ο, το, το πού γίνεται η φορολογία στις διεθνείς μεταφορές η ισχύουσα κατάσταση σημαίνει ότι δύο χώρες φορολογούσαν το ίδιο σημείο και αυτό δεν είναι εύκολο. Όταν δημιουργήθηκε η εσωτερική αγορά η Επιτροπή, το 1992 ήδη είχε κάνει μία πρόταση λέγοντας ότι η φορολογία θα γίνει στο σημείο αναχώρησης. Αλλά τα κράτη-μέλη έχουν επιλογή. Αυτό ζητά το ίδιο. Δυστυχώ η Επιτροπή δεν μπορούσε να περάσει την πρότασή τη το 1992. Έκτοτε λειτουργεί ένα μεταβατικό σύστημα ΦΠΑ, όχι οριστικό, διότι ούτε και οι συντελεστέ ήταν οι ίδιοι, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για κοινού κανόνε στα κράτη-μέλη. Υπήρχαν πολλέ παρεκκλήσει προ εξαιρέσει για να φτάσουμε σε κάποια ελάχιστα όρια για την εσωτερική αγορά. Η Κομισιόν έχει προτείνει κανόνε για αυτό το οριστικό σύστημα. Δυστυχώ, τόσο όχι δυστυχώ, αυτό είναι τεράστιο εγχείρημα. Η πρόταση περιορίστηκε στην παροχή αγαθών, στην μεταβίβαση αγαθών. Δεν υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες ε, προτάσεις για τις υπηρεσίες όπως τις μεταφορές. Αυτό δεν έγινε. Αναγγέλθηκε σε μια ανακοίνωση προς, ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνέχεια του προγράμματος της Επιτροπής για το θέμα αυτό. Αυτά μπορώ να σας πούμε προς το παρόν. Τώρα, γιατί δεν έχει προχωρήσει η πρόταση για τις υπηρεσίες, ε, να σας πω ότι είναι πολύ σύνθετη. Γενικά, οι κοινοί κανόνες για το ΦΠΑ, για τις υπηρεσίες, ωστόσο, ιδίως στις οδομικές μεταφορές, υπάρχει μία εξαίρεση. Για τα αγαθά χρειάζεται μεγαλύτερη ε, ανάγκη Δεν θέλω να μπω σε τεχνικά θέματα. Αυτά. Ευχαριστούμε. Ο κ. Βίντσι για τις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι οι εξηγήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευσταθούν. Είναι καλές. Αυτή τη γραμμή να ακολουθήσουμε πρέπει. Ο ΦΠΑ είναι εθνική αρμοδιότης κυρίως. Καλό να υπάρχει η σύσταση και ευελιξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ούτω ώστε να επιτρέπεται στα κράτη-μέλη η επιλογή. Μπορεί να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, διότι οι δημόσιες μεταφορές, οι μαζικές μεταφορές ανήκουν στην Πράσινη Συμφωνία. Και όλες οι αναφορές που συζητήσαμε έχουν κάποια σχέση με την Πράσινη Συμφωνία. Θα χρειαστούμε ευελιξία στο τομέα αυτό. Έχουμε και τον φόρο καυσίμων στις αερομεταφορές που ακολουθήσουμε και προσέγγιση ΦΠΑ. Ας παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ίσως έχουμε και την γνωμοδότηση της Αρμόδιας Επιτροπής, της Ήτρα νομίζω. Α, τραν, τραν. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άουκεν. Οι, πράσινοι συμφωνούν με τους αναφέροντες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις για να συμβεί αυτό. Ίσως να ετοιμάσουμε και ακρόαση. Uh, Έχουμε πρόβλημα με τις σιδηροδρομικές μεταφορές κυρίως στην Ευρώπη. Μαζί με την Τράμπο διοργανώσουμε ε, μια ακρόαση πάνω σε αυτό. Βεβαίως να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Τέλεια. Έχοντας ακούσει όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, προτείνω να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά και να ζητήσουμε ενημέρωση για τις πληροφορίες από την Κομισιόν, ιδίως για την πορεία της νομοθεσίας για το ΦΠΑ είπε η Επιτροπή τον Ιανουάριο δεν θα αξιολογηθεί στο Συμβούλιο η πρόταση του 2018 από την Επιτροπή, αλλά ίσως αυτό να είναι ένα σημαντικό σημείο για τις μεταφορές. Ό,τι αφορά την πρόταση, το βλέπουμε και με τους συντονιστές, παραμένει ανοιχτή η αναφορά σε κάθε περίπτωση. Επόμενο θέμα 274 του 2019 αναφορά ενός Φιλανδού πολίτη για την φορολογία ηλεκτρικών ε, αυτοκινήτων που φορτίζουν στην Φιλανδία. Λείπει αναφέρον. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το λόγο. Δύο μέλη, της Κομισιόν δηλαδή. Ο κύριος Τουομίνεν από την Γενική Διεύθυνση Ταξούντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η αναφορά περιέχει δύο διαφορετικές πτυχές. Ασχολείται με άμεση και έμεση φορολόγηση. Κάποια σχόλια θα κάνω για το ένα και ο συνάδελφος για το άλλο. Καταγγέλει τη νέα νομοθεσία της Φιλανδίας, ο αναφέρον. Σύμφωνα με αυτή, η φόρτιση στο χώρο εργασίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων με κόστος του εργοδότη είναι ε, κάτι που θα πρέπει να φερείται ως όφελος από, την φορολογική δήλωση ως όφελος που έχει ο εργαζόμενος. Αυτό ταιριάζει και με άλλα πλεονεκτήματα που δίνει μια εταιρεία, παραδείγματο χάρη, βάτσες για γεύματα, δωρεάν τηλεφωνήματα, ε, εταιρικό αυτοκίνητο κλπ. Εδώ δεν έχουμε δευτερογενή νομοθεσία τη Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Αρμοδιότητες βασικά είναι των κρατών μελών το πώς αντιμετωπίζουν το θέμα. Και η Φιλανδία αποφάσισε τούτο τρόπος 30 ευρώ να φορολογήσει αυτό το όφελο το μήνα και προστίθεται στο φορολογούμενο <clears throat> ε, εισόδημα του φορολογούμενου. Δεν έχει διασυνοριακή διάσταση αυτό το μέτρο. Δεν, υπάρχει διάκριση βάση ε, ή τόπου διαμονής. Άρα οι δυνατότητες παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ανύπαρκτες. Αρκετά για τον άμεσο φόρο θα μιλήσει τώρα ο συνάδελφος για το άλλο θέμα. Ή συνάδελφος. Ο αναφέρον ανέφερε κάτι άλλο. για φορολόγηση φυσικού αερίου και δίζελ. Για τα ιδιοταχή δεν υπάρχει εναρμόνιση όσον αφορά δίζελ ή βενζίνη. Έχουν αποτύχει οι προτάσεις μας. Τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα να φορολογήσουν για τέλη κυκλοφορίας, τέλη πινακίδων κλπ. Αν δεν υπάρχει διάκριση άμεση έμεση προϊόντων που προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη. Εδώ δεν βλέπουμε να υπάρχει διάκριση στη Φιλανδία. Σχετικά με τη φορολόγηση των καυσίμων, έχουμε την οδηγία για τον ενεργειακό φόρο, καθορίζεται η ελάχιστη φορολόγηση διάφορων καψίμων και σαν τμήμα της Πράσινης Συμφωνίας εξετάζεται μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα υποβληθεί το επόμενο καλοκαίρι το 2020. Βάσει αυτού δεν βλέπουμε να υπάρχει παραβίαση του ενωσιακού δικαίου άρα δεν πάει καν τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Γιάρη, κύριε Άουκεν. Δεν ξέρω, λέει κύριε Γιάρη. Δεν ξέρω πώς οι δυο μας μπορούμε να τα βρούμε εδώ με την κυρία Άουκεν. Εγώ έχω ε, ανάμεικτα συναισθήματα, τα ίδια επιχειρήματα ε, ή μάλλον ίδιο αριθμό επιχειρημάτων για να μην είναι ανοιχτή να κλείσει αναφορά, αλλά μάλλον θα έλεγα να κλείσει. Δεν ξέρω τι λέει η κυρία Άουκεν. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει και αυτή να πει την άποψή της. Ε, θα σας ακούσω, ε. μόνο αυτή τη φορά θα σας ακούσω όμως. Ε. Πάρα πολύ είναι εθνική νομοθεσία και δεν θα ήθελα να παρέμβει η γερμανική μηχανία για τη φορολόγηση της βενζίνης η Δανία για παράδειγμα. Αν μείνει ε, μέσα στην πρόθεση του Πράσινου Συμφώνου, την από θα μπορούσε να παραμείνει ανοιχτή. Γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάμε την πράσινη φορολογία αλλά και εγώ έχω τις αμφιβολίες μου. Λοιπόν, πρόεδρος, η δική μου πρόταση είναι να κλείσει η αναφορά. Άκουσα την Κομισιόν, δεν έχει αρμοδιότητα λέει, αλλά είναι εθνική αρμοδιότητα, άρα για τη Φιλανδία πρόκειται και αφού μας λέει ότι δεν υπάρχει φορολογική διακριτική μεταρρύθμιση, ε, μεταχείριση ε, καθότι πρόκειται για εσωτερικό φορολογικό ζήτημα, ε, να κλείσει. Τώρα δεν ξέρω άποψη των κυρίων, του κύριου Γιάννη και της κυρίας Άκερ να παραμείνει ανοιχτή για να δούμε τα της ενέργειας που θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα η νέα Κομισιόν ή έχουμε και τον νέο παράσινο σύμφωνο αυτή την νομοθεσία να μην είναι ανοιχτή ή να κλείσει. Συμφωνείτε να κλείσει. Α, όχι, ανοιχτή. Λέει κυρία Όκεν. Μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο, ή μάλλον η Νέα επιτροπη για την φορολογία. Άρα λέει ο κύριο Γιάρα, όχι στο δίνεκε ανοιχτή, αλλά περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις για τη φορολογία. Είδατε, να τα βρήκαμε κυρία Όκεν, συμφωνήσαμε σήμερα οι δυο μα. Πρόεδρος, ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με την οδηγία για τη φορολόγηση και για το πράσινο σύμφωνο. Πάμε στο 10, έχει κατόπιν αιτήματος ε, του αναφέροντος αναβληθεί, οπότε περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης ε, που είναι η δική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. 14, παρθμό 14 του 2019. Είμαστε αυτή η η κυρία Τάρτερ, στο βήμα. Δέκα λεπτάκια, ανεμή, για να μας παρουσιάσετε την έκθεση αυτή. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες ε, διαβουλεύσεις.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 Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την, ε, ότι οι διαβουλεύσεις κομισιών εντάσσουν τους πολίτες αλλά δεν καλύπτουν ε, τα πάντα. Ε, η, το Ελεκτικό Συνέδριο πήρε το αίτημα από εσά για να δώσουμε μία, για κάνουμε μία μελέτη για το πώς η Επιτροπή εμπλέκει τους πολίτες. Ε, ο στόχος να ζητήσουμε την άποψη των πολιτών και την... να δούμε πώς λειτουργεί το εργαλείο αυτό της Επιτροπής. Ξεκινώ προσπαθώντας δεν δουλεύει πρώτα πρώτα γιατί κάναμε την μελέτη, ποιος είναι ο στόχος της και να παρουσιάσω τα ευρήματα και τις συστάσεις. Γιατί κάναμε αυτό, αυτή τη μελέτη. Πρώτα πρώτα, υπάρχει το άρθρο 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση με, που δίνει στην Επιτροπή την υποχρέωση να διαβουλεύεται με τους πολίτες και τις ενώσεις πολιτών σε όλους τους τομείς δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή πρέπει να κάνει ευρεία διαβούλευση δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς να εμπλακούν στην διαμόρφωση της πολιτικής. Υπάρχει και η Λευκή Επίβλος για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση του 2001, όπου η Επιτροπή δεσμεύθηκε να έρθει σε επαφή με πολίτες και εμπλεκόμενους. Υπάρχει και η δική μας στρατηγική του Ενεκτικού Συνεδρίου για την περίοδο 18-20 και βεβαίως το αίτημα της Επιτροπής ΠΕΤΗ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αξιολογήσουμε το πώς οι πολίτες μπορούν να μετάσχουν απευθείας στην διαμόρφωση, της, στην ομοπαρασκευαστική διαδικασία της Ένωσης. Ποιος ήταν ο στόχος του, της μελέτης να δούμε κατά πόσον οι, οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι αποτελεσματικές και καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τους πολίτες χρησιμοποιώντας την συμβολή τους. Αξιολογήσαμε κατά πόσον ο σχεδιασμός του πλαισίου της Επιτροπής για τις, διαμούσεις, για τις δημόσιες διαβουλεύσεις αντικατοπτρίζει σωστή πρακτική, αν η Επιτροπή προετοίμασε και επικοινώνησε με τους ε, πολίτες ούτως ώστε να συμμετάσχουν αυτοί με εύκολο τρόπο και αν ανάλυσε τα στοιχεία, τα, τα στοιχεία που αναλύονται είναι εύλογα και κατανοητά, καθώς και το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Κατά μέσο πρέπει να πούμε ότι η Επιτροπή κάνει πάνω από 100 δημόσιες διαβουλεύσεις κάθε χρόνο. Αναλύσαμε 26 δημόσιες διαβουλεύσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2016 και 2018 με 5, από 5 γενικές διευθύνσεις βάσει των διαβουλεύσεων ο έλεγχο είχε περιλαμβάνει συνεντεύξεις με το προσωπικό, με τα κρατημέλη και με τον ΩΣΑ, εξετάζοντα βασικά κείμενα και εμπλεκόμενων φορέων και ε, με διαβούλευση ομάδας εμπειρογνωμών. Επίση κάναμε μία μελέτη κατανόηση μεταξύ 6.000 πολιτών που μετήχαν στο δείγμα μα για να συμπληρώσουμε τα ευρήματά μας. Πήραμε πάνω από 2.200 απαντήσεις από τους 6.000 αυτούς ανθρώπους. Τι βρήκαμε. Πρώτον, το πλαίσιο της Επιτροπής για τις δημόσιες διαβουλεύσεις ορίζεται από, το, ε, από την εργαλειοθήκη για την καλύτερη νομοθεσία με συγκεκριμένες καθοδητήριες γραμμές όπως υιοθετήθηκαν το 2015. Τον Ιούλιο του 2017 η Επιτροπή υιοθέτησε και ένα πρόσθετο πλέγμα διαβουλε... οδηγιών για το πώς διαβουλεύεται με τους πολίτες. Με βάση τις 26 διαβουλεύσεις που εξετάσαμε και την δική μας perception survey, βρήκαμε ότι περίπου τα δύο τρίτα των, των απαντήσεων έδειχναν ικανοποίηση με τη διαδικασία διαβούλευσης. Το υψηλό επίπεδο των ε, ε, ε, των προτάσεων της Επιτροπής έγινε ε, δεκτό και από τον ΩΣΑ. Είναι πρώτη στην εμπλοκή των πολιτών στις χώρες ΩΣΑ. Υπήρχαν ελλείψεις τόσο σε ό,τι φορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της δημόσιας διαβούλευσης που θα εξηγήσω κατόπιν. Τι βρήκαμε. Πρώτα πρώτα. Αν δείτε αυτό το γράφημα δεξιά διαπιστώνετε ότι υπάρχει χαμηλή δυνατότητα πρόσβασης. Πολλές δημόσιες διαβουλεύσεις ε, έχουν 22, 24, 27, 441 άτομα που μετήχαν. Μόνο οι τελευταίες μεγάλες ε, έχουν ε, ε, σημασία ότι η τελευταία είναι για το αν θα έχουμε το θερινό, θερινή ή χειμερινή ώρα, την ξέρετε όλοι. Όλα τα άλλα είχαν μικρή πρόσβαση στους πολίτες, αν λάβουμε υπόψη ότι στην Ευρώπη έχουμε μισό, εκατο, μισό δισεκατομμύριο πολιτών. Το να έχουμε τώρα 70, 100, 200 απαντήσεις δεν είναι καλό. Δεν υπήρχε λοιπόν στρατηγική διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση είναι κομμάτι μιας ευρείας διαδικασίας. Δεν ξέρουμε ποια εργαλεία χρησιμοποιεί η Επιτροπή ποιο εργαλείο συμπληρώνει άλλο εργαλείο. Για πολύ τεχνικά θέματα δεν είναι εύλογο να υπάρχει διαβούλευση του γενικού κοινού. Επίσης, υπήρχαν προβλήματα σε ό,τι αφορά τη χρήση γλώσσας. Κάποια ερωτηματολόγια ήταν πολύ μεγάλα, πολύ, πολύ σύνθετα. Κάποια ερωτηματολόγια δεν ήταν μεταφρασμένα σε άλλες γλώσσες, αλλά μόνο στα αγγλικά. Κάτι που για πολλούς πολίτες βέβαια δεν είναι εύκολο. Το χρονοδιάγραμμα τώρα, 92% των διαφυλεύσεων σεβάστηκαν το, τις 12 εβδομάδες για, το, για τις απαντήσεις, αλλά δεν, ε, κάποιοι μας είπαν ότι δεν είχαν χρόνο να απαντήσουν σε κάποιες. Υπήρχαν κάποια, κάποια προβλήματα και στην παρακολούθηση και στο monitoring δηλαδή και στην αξιολόγηση. Τι βρήκαμε. Αυτό είναι το slide για, το, τη χειμερινή ώρα. Ε, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μεγάλη γεωγραφική ανισότητα. Οι περισσότεροι από αυτούς που απάντησαν ήταν Γερμανοί και Αυστριακοί. Αν δείτε τα χρώματα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας μεταξύ νότου-βορρά. Δηλαδή νότου, κέντρου και βορράς. Και βορρά. Η Γερμανία και η Αυστρία είναι τα βυσινή χρώματα. Τώρα δεξιά στο γράφημα θα δείτε ότι 40% των απαντήσεων δόθηκαν στις δύο τελευταίες μέρες της διαβούλευσης. Παροχή πληροφοριών για την δραστηριότητα ε, της διαβούλευσης. Εδώ υπήρχαν κενά και στην επεξεργασία των δεδομένων και στην ανάλυση των δεδομένων δεν, υπήρχαν, ε, δεν υπήρχε το feedback προς αυτούς που μετήχαν και με περιορισμένη δημοσιότητα. Οι άνθρωποι στην έκθεση λένε είναι ικανοποιημένοι που ζητά την άποψή τους η Επιτροπή, αλλά από την άλλη δεν είναι ικανοποιημένοι γιατί δεν παίρνουν feedback. τέλος πάντων δεν μαθαίνουν τι έγινε μετά. Προχωρώντας, δεύτερη σύσταση. το, frame, το πλαίσιο της Επιτροπής. Η πρώτη, μας η πρώτη σύσταση είναι η Επιτροπή να παρακολουθεί καλύτερα τη δημόσια διαβούλευση, βελτιώνοντας τις ε, οδηγίες με συγκεκριμένους δείκτες που πρέπει να παρακολουθηθούν και να γίνει αναφορά σε αυτούς και ταυτόχρονα συστηματική αξιολόγηση του κατά πόσο η δημόσια διαβούλευση πέτυχε τους στόχους της. Παλεύω λίγο εδώ με το PowerPoint, αλλά προχωράω. Όχι, πρέπει να πάω πίσω, συγγνώμη, με συγχωρείτε, τα Δεύτερη σύσταση. Στρατηγική διαβούλευση. Να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών. Και για να γίνει αυτό, το πρέπει να εξηγήσει ποιε δραστηριότητε διαβούλευση επιλέγει για ποια δραστηριότητα. Εμεί στην έκθεσή μα δίνουμε ένα γράφημα που λέμε δεν πρέπει να έχουμε μόνο online αλλά συναντήσει αντιπροσωπευτική δημοκρατία στο κοινοβούλιο. Κάθε επίπεδο πρέπει να συμπληρώνει τα άλλα. Δηλαδή η διαβούλευση δεν είναι καλή μόνο με τρει ανθρώπου που απαντάνε. Διαβούλευση ούτε είναι σωστή μια διαβούλευση που είναι μόνο συνάντηση εμπλεκομένων φορέων. Επίσης να διευκρινίσουμε ότι καλό θα ήταν να μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες τα ερωτηματολόγια να προσαρμόσουμε τα μέτρα επικοινωνίας. Τι κάνεις όταν έχεις μία απάντηση από 500 πολίτες. Πώς μπορείς να καλύψεις το κενό μεταξύ του ευρωπαϊκού έργου και των 500 ή των, περισσότερων πολιτών. Πώς μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία αν έχει μία απάντηση 500 ανθρώπων από τα 500 εκατομμύρια. Τι αντλείς από αυτό δηλαδή. Άρα, με, πρέπει να εμπλέκουμε τι αντιπροσωπείες τη στα κράτη-μέλη περισσότερο. Τέταρτο, τέταρτη σύσταση. Τα γλωσσικά. Είπα ότι κάποια κείμενα δεν είχαν μεταφραθεί, ήταν μόνο στα αγγλικά. Αυτό δυσκολεύει κάποια κράτη-μέλη, πολλού πολίτες. Πρέπει οι διαβουλεύσει να βασίζονται σε γενικέ εποπτείε για, το, για τους πολίτες. Σύσταση 5. Κάτι πολύ σημαντικό είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τη διαδικασία διαβούλευσης από τη χειραγώγηση. Για να γίνει αυτό πρέπει η Επιτροπή να έχει υψηλότερα επίπεδα επεξεργασίας δεδομένων. Αυτή τη στιγμή τα συστήματα δεν είναι επαρκώς προστατευμένα. Δεν είναι σαφές κατά πόσον οι απαντήσεις των ανθρώπων μπορεί να έρχονται από την Ευρώπη, αλλά μπορεί να έρχονται και από εκτός Ευρώπης. Μπορεί ένα άτομο να έχει μετάσχει περισσότερο από μία φορά. Ξέρω ότι δουλεύει σκληρά στον τομέα αυτό για την επεξεργασία δεδομένων η Επιτροπή, αλλά να το παλέψει ακόμα περισσότερο. Τελευταία σύσταση. Feedback. Είπαμε, ο κόσμο είναι ευχαριστημένο που ζητάνε την άποψή του, αλλά δεν έχουν ενημέρωση τι έγινε μετά. Δεν ξέρουν αν η συμβολή του λήφθηκε υπόψη ή όχι. Αυτό είναι, Αυτά είναι τα βασικά σημεία της έκθεσής μας. Περιμένω με ανεπομονησία τις ερωτήσεις σας. Ελπίζω το έγγραφο αυτό να συμβάλλει στην βελτίωση των εργασιών της Επιτροπής ΠΕΤΗ. Υπάρχει χώρος για βελτίωση, πρόκειται για καλές πρωτοβουλίες αυτές της Κομισιόν. Μπράβο στην Κομισιόν που πάει και ρωτάει τους πολίτες. Πάντα μπορούμε να βελτιωθούμε, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ. Um, Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει πρόεδρος mm. Αντωνίνα Τσιπολόνη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ το Ελληνικό Συνέδριο για αυτή την πολύ καλή έκθεση. Χαρήκαμε που τη λάβαμε. Δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά κάνει τη διαβούλευση με τους πολίτες. Εν γέννη το σύστημα θεωρείται καλό, το αναγνωρίζει και όσα το σημαντικότερο είναι ότι αναγνωρίζουν οι πολίτες, διότι αυτοί που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις ε, αυξάνονται. Έχουν τετραπλασιαστεί οι συμμετέχοντες. Και είναι θετική ανταπόκριση, η άποψη για το σύστημά μας και αυξάνεται η εμπιστοσύνη τους. Ενθαρρυντικά αυτά. Συμφωνούμε όμως ότι κάποιες βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε. Κάναμε και εμείς μια αποτίμηση στα πέσεις πολιτικής για καλύτερη ε, θέσπιση νομοθεσίας και είδαμε κάποια στοιχεία που αναφέρει και το ελεκτικό συνέδριο. Πρέπει να πλησιάσουν περισσότερους, να βελτιωθεί η ποιότητα των διαβουλεύσεων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη προστασία των δεδομένων. Ταυτόχρονα να δίνεται μια σωστή συνέχεια στις διαβουλεύσεις. Θέλουμε να αλλάξουμε δεόντως το σύστημα. Να συμμορφωθούμε με τις συστάσεις. Τις δεχτήκαμε όλες. Θετικότατη συνεισφορά στην ανάπτυξη της ατζέντα μας για την καλύτερη νομοθεσία που θα επιδιώξουμε και θέλουμε την δυνα... τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση με τους πολίτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Άουκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, Υπάρχουν περιθώρια βελτίωση από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό το θέμα της θερινής ώρας κανείς δεν το έχει ακούσει στη Δανία. Και εκείνοι που έδωσαν απάντηση είναι αυτοί που είναι πολύ δραστηριοποιημένοι στο θέμα. Μετά μου μίλησε κάποια αθλητική οργάνωση και είχαν στενοχωρηθεί γιατί θα χάνανε τη μία, με την αλλαγή της ώρας θα χάνανε μία ώρα άθλησης. Και τους είπα, «Ε, δεν μου το είπατε έγκαιρα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε σωστή χρήση του μέσου. Να την ξέρει και ο κόσμος ότι υπάρχει. Πόσους έχετε στη Γερμανία, Πίτερ, τι είπες? Αρκετούς, ε αλλά είναι πολύ μικρός αριθμός σε συγκρίση με όλους τους ε, κατοίκους. Στην Επιτροπή Αναφορών είδαμε ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στις εργασίες του Συμβουλίου. Αν μπορούσαμε να παρακολουθούμε και τις δύο πτυχές της θέσης της νομοθεσίας τα εθνικά κοινοβούλια και εθνικός τύπος να μπορεί να δει τι γίνεται στα κοινοβούλια. Τότε το εργαλείο μας ε, για τη συμμετοχή των πολιτών θα ήταν αποτελεσματικότερο. Αν ήταν πιο γνωστό στους πολίτες τι κάνει η κυβέρνησή τους. Δεν ξέρουν πώς δουλεύουν οι ομάδες εργασίας, οι επιτροπές εργασίας κλπ, οι πολίτες. Είχαμε έκθεση το 2018 του συνηγόρου του πολίτη και Επιτροπή ΑΦΚΟ και Αναφορών Πέρσι έδωσε κάποια σχετική ε, γνωμοδότηση που υποστήριζαν το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τις συστάσεις της εκθέσεως του συνηγόρου του πολίτη. Εάν δεν παρακολουθεί κανείς τα τεκτενόμενα βλέπει ότι δεν υπάρχουν καταστοιχεία για την εξοικονόμηση ενεργείας με την αλλαγή της ώρας. Δεν έχουμε στοιχεία. Άλλα λένε, άλλα στοιχεία υπάρχουν. Στην Φιλανδία το καλοκαίρι δεν, δίνει, δεν δει καθόλου ήλιος. Άρα είναι μπελάς να αλλάζει την ώρα. Στο Όσλο τους αρέσει. Εκεί κάνει τη διαφορά η αλλαγή της ώρας. Πρέπει να δίνουμε σαφέστερα τα στοιχεία. Κάνουμε εμείς ακροάσεις, ακούμε πυρογνώμονες, εξετάζουμε στοιχεία κλπ. αλλά κόσμος δεν ξέρει. Και πώς θα πειραζόταν όλοι. Εμείς αλλάζουμε... Ε, ε, εάν βασιζόμαστε στα στοιχεία, εμεί που ταξιδεύουμε ψυχνά δύο φορέ την εβδομάδα θα ήμασταν άρρωστοι, γιατί έτσι διατηνόταν κάποιε εκθέσει και στοιχεία. Μεροληπτική ήταν η προσέγγιση κατά την απόψη μου αφορά ώρα. Εμένα μου αρέσει, μου αρέσει και αυτό είναι πρόβλημα. Μου αρέσει τερινή ώρα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και δεν είχα και προβλήματα όταν είχα μικρά παιδιά, προσαρμόστηκα άνετα στην αλλαγή της ώρας. Πρέπει να έχουμε σωστή βάση για τη συμμετοχή των πολιτών. Στο άρθρο 1 και στο 10 νομίζω ότι αναφέρεται ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα συμμετοχή στη δημοκρατία με τον στενότερο και διαφανέστερο τρόπο. Αν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν να τι κάνει η κυβέρνησή τους, τι θα κάνουν οι πολίτες. Δεν έχουν καμία τύχη και του ρωτάμε τι σκέφτεσαι για αυτό, τι σκέφτεσαι για εκείνο και άντε να σε ακούσει κανεί. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα καλύτερα αποτελέσματα τα είχαμε θερινή ώρα. Γι' αυτό ήταν σκανδαλώδες τα λέω εγώ. Θα διαβάσω την έκθεση. Να προσθέσετε και το αίτημα το μεγάλο του Κοινοβουλίου και του συνηγόρου του πολίτη. να κινηθούν και κυβερνήσεις. Δεν είναι διακυβερνητικό φορέας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο κινούμαστε εμείς από τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι διπλωμάτες. Στους διπλωμάτες δεν του αρέσει καθόλου η διαφάνεια δυστυχώ. Κύριε ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη. καταρχά. και για την ε, σύντομη, ίσως όχι και τόσο ίσως ε, οργανωμένη θα ήθελα να πω ε, παρουσίαση, προφορική παρουσίαση. Υπάρχει δημοκρατία στην Ευρώπη για να είμαστε closer to the people, πιο κοντά στον πολίτη και σίγουρα αυτές οι δημόσιες διαβουλεύσεις είναι ένα πάρα πολύτιμο, πολύ, πολύτιμο εργαλείο για αυτό. Συμφωνώ ότι είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε και θέλουμε. Είναι πραγματικά καλό να προβάλλουμε τις ε, διάφορες προτάσεις νομοθεσίας προτού γίνουν νομοθεσία. Ε, είναι σημαντικό να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό. Βέβαια θα πρέπει και η γλώσσα ε, να είναι κατανοητή ε, και Επομένως, να μην γίνονται οι εκδόσεις μόνο σε τρεις γλώσσες ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θέλουμε να υπάρχει προβολή και αν θέλουμε να υπάρχει διαβούλευση, θα πρέπει να μπορεί ο πολίτης να καταλάβει. Και επίσης δεν θα πρέπει αυτές οι εκδόσεις ή όλες αυτές οι δημοσιεύσεις να είναι για λίγους, ε, αλλά για τον πολίτη. Δηλαδή όχι για ομάδες συμφερόντων ή για κάποιους ε, συγκεκριμένους κύκλους, αλλά να είναι διαθέσιμες και κατανοητές ε, από το πλατή κοινό. Και επίσης ε, βλέπουμε και τις ομάδες ε, επισκεπτών. Πάρα πολύ λίγοι τα γνωρίζουν. Πολύ λίγοι γνωρίζουν για τις προτάσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Φανταστείτε αν μπορεί κάποιος πολίτης ε, να συνεισφέρει, δηλαδή εκφράζοντας και την άποψή του για κάποιες προτάσεις νομοθεσίας. Αλλά δυστυχώς είναι άγνωστα όλα αυτά στους περισσότερους. Επίσης, πράγματι δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χειραγώγηση. Συμφωνώ και σε αυτό και σε ό,τι αφορά το feedback. Ε, εγώ σας ρωτώ, ε, έχουμε ας πούμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί πάρα πολύ ε, και έχουμε πάρα πολλούς ε, που απαντάνε. Τι θα λέμε, ευχαριστούμε πολύ για το feedback ε, ή ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Εγώ σας γυρίζω το ερώτημα πώς θα κάνουμε τον κόσμο να θέλει να ενδιαφερθεί και να συμμετάσχει περισσότερο. Οι δημόσιες αυτές λοιπόν διαβουλεύσεις είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για την δημοκρατία και για την λαϊκή συμμετοχή. Δυστυχώς όμως είναι κάτι πάρα πολύ λίγο γνωστό και ελπίζω η δική σας η μελέτη να μπορέσει να συνεισφέρει ε, στο να έχουμε και νέες ιδέες ε, που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Όχι δηλαδή να έχουμε άσκηση κριτικής ε, σε ένα νομοθέτημα, αφότου πλέον αυτό έχει ε, οριστικοποιηθεί, αλλά να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών εκ των προτέρων από την αρχή. Νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε στον περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Ε, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά ε, το Ελεκτικό Συνέδριο για την έκθεση και για τα όσα μας ε, μεταφέρατε που θα μας επιτρέψουν, πιστεύω, να βελτιώσουμε Γιατί πραγματικά είναι περίεργο και ενίοτε λυπηρό το ότι υπάρχει τόσο λίγη συμμετοχή στι δημόσιε αυτέ διαβουλεύσει από πλευρά τη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση. Εγώ προέρχομαι ε, από ένα κράτος ε, μέλος που ε, επίσης δεν έχουμε καλά αποτελέσματα με την έννοια ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν πώς, πού, σε ποια ιστοσελίδα να μπω, σε ποια γλώσσα να συνδεθώ. Πολλές φορές μπορεί να είναι μόνο στα αγγλικά και όχι στις 27 γλώσσες, ε, μάλλον στις γλώσσες των 27 κρατών μελών. Είμαστε στον 21ο αιώνα, πρέπει να προσαρμοστούμε ε, και σε ό,τι αφορά τα μίντια και να προσεγγίσουμε τους πολίτες. Πού που βρίσκονται οι πολίτες, βρίσκονται στα κοινωνικά δίκτυα ή επίσης ε, μπροστά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο. Ε, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι όταν εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι ακούν ραδιόφωνο και πρέπει και εκεί να μπορέσουμε να αυξήσουμε την προβολή. Και αυτό που είπατε για την ε, ώρα, τη θερινή, τη χειμερινή, είδαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή εκεί, άρα πρέπει να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών. Θέλω να συγχαρώ την ε, Επιτροπή μας που είχε αυτή την πρωτοβουλία να αναθέσει αυτή την έκθεση στη, στο Ελληνικό Συνέδριο για να έρθει εδώ και να μας παρουσιάσει ε, το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις δημόσιες διαβουλεύσεις που είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Πρέπει να είναι σίγουρα ε, πιο μεγάλη η προβολή, η διαφάνεια και πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στις δημόσιες αυτές διαβουλεύσεις. Θέλουμε λοιπόν η Κομισιόν να αναζητήσει τους πολίτες εκεί όπου βρίσκονται. Δεν είναι πίσω από την επίσημη ευρωπαϊκή εφημερίδα οι πολίτες, αλλά είναι στο σπίτι τους, ε, στο δίκτυο, στην οθόνη, ε, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Εκεί πρέπει να γίνονται και αυτές οι δημόσιες Σε Ευχαριστώ πάντως για την πολύ καλή δουλειά, γιατί νομίζω ότι αυτό θα βελτιώσει ε, την δυνατότητα επαφή των θεσμικών οργάνων με του πολίτε. Σα ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε, αν συμφωνείτε τώρα, στο επόμενο σημείο της μερισιάς διάταξης, το υπαριθμόν 1296, υπαριθμόν αναφορά, ισπανική Ιθαγένειας. ο αναφέρον. Είναι εδώ αναφέρον, ε, θα μας ε, μιλήσει για τη δημιουργία ενός πρότυπου σε ό,τι αφορά την ε, ατμοσφαιρική ρήπανση και την ταξινόμηση των οχημάτων για διάφορες ε, περιορισμούς στην οδική κυκλοφορία. Οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρουν τι ανησυχίε που περιέχει αναφορά. Να επαναλάβω καταρχήν ότι οδηγεί το περιβάλλον και την ποιότητα του σφαιρικού αέρα λέει ότι θα εξασφαλίσει κάτι μέλη ότι οι συγκεντρώσει ρηπαντών στην ατμόσφαιρα δεν ξεπερνούν τις οριακέ τιμές που καθορίζουν την οδηγία. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών υποχρεώνονται κράτη-μέλη να, βάλουν, να εφαρμόσουν σχέδια και κατάλληλα μέτρα, ούτω ώστε η περίοδο υπέρβαση να είναι η βραχύτερη δυνατή. Η επιλογή των μέτρων εξαρτάται τι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να επιβαληθεί μέσω του κανονισμού για περιορισμό κυκλοφορία των οχημάτων, όπω και ζώνε με χαμηλή εκπομπή. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε και θεωρούμε ότι οι πληροφορίες και η παροχή πληροφοριών δυνάμει του κανονισμού μπορεί να βελτιωθούν για να διευκολυνθεί η κατάσταση για του οδηγού πληροφορίες που χορηγούνται σε αυτό το πλαίσιο. Ο κανόνας για μια ψηφιακή πύλη επιβάλλει οι δημόσιε να δίνουν στο διαδίκτυο και στου πολίτε και σε επιχειρήσει δεδομένα για το εφαρμοστέους κανόνες εθνικό ή τοπικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο και στου δικού χρήστες να δίνονται πληροφορίες. Και αυτό να γίνεται μέχρι το τέλος του 2020. Να βρίσκονται εύκολα οι πληροφορίες, να είναι εύληπτε. και μέχρι το 2023 τα κράτη-μέλη θα επιτρέπουν να μπορούν να πάρουν ετικέτες για εκπομπέ, ε, να κάνουν την αίτηση στο διαδίκτυο οι οδηγοί και να μπορούν να πάρουν το αυτοκόλλητο. Θα γίνουν και άλλες αλλαγές στα μέτρα. και δεν ε, ξέρουμε δεν, ε, από ό,τι θα δημοσιευθούν οι κατάλληλε πληροφορίε σε μελλοντικά έγγραφα θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Θέλουμε να εφαρμόσουμε το 2020 ένα σχέδιο για ευφύ κινητικότητα στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας. Εξετάζουμε το θέμα και αξιολογώντας και το πακέτο για νηστική κινητικότητα του 2013. Εκεί θα δούμε ποια είναι η πολιτική που χρησιμοποιείται στις ε, πόλεις και η νομοθεσία για τα οχήματα και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Άλλη εξέλιξη. Μετά την απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση. Το αναφερειμένο σχέδιο κατευθύνες γραμμές για την αστική κινητικότητα ε, έχουν δημοσιευτεί κανόνες και ένα σχετικό έγγραφο για, που αφορά τους κανονισμούς που ισχύουν για την κινητικότητα της πόλης. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει δώσει χρηματοδότηση για παρασκευαστική δράση του Ευρωκοινοβουλίου για να παρέχονται πληροφορίες στους οδηγούς που είναι εύχριστες. Χρειάζεται τυποποίηση και παροχή δεδομένων. Όπως να δίνονται πληροφορίες σε συσκευές πλοήγησης και στις εφαρμογές πρέπει να παράγονται πιο εύκολα πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό περί ενίας ε, ψηφιακής πύλης. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάρ. Νομίζω ότι έχει ήρθει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα να φέρουν αν συνεχίσουμε έτσι με αυτές τις διαφορετικές ταξινομήσεις και με τις ε, διαφορετικές ε, ζώνες ε, κυκλοφορίας για την ταξινόμηση χημάτων, τα περιβαλλοντικές τα κτλ. Πράγματι θέλουμε να έχουμε εσωτερική αγορά και ελευθερία κυκλοφορίας. Αλλιώς θα τα καταστρέψουμε. Εγώ έχω πρόβλημα ήδη να καταλάω ίσο το γερμανικό σύστημα και είμαι Γερμανός. Ε, εντάξει, υπάρχει ένα ε, αυτοκόλλητο που μπορούμε να το ε, κολλήσουμε, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αποκλείονται κάποιοι δρόμοι, αν υπάρχει παραδείγματος χάρη ε, κάποιο καιρό φαινόμενο. Ε, και φαντάζομαι ότι και για την ε, Ελλάδα πρέπει οι άλλες πολύ ωραίες περιοχές που θέλουμε να επισκεφθούμε, να μπαίνουν κάποιες πινακίδες ε, αλλά δεν είναι εύκολο να καταλαβαίνει κανείς. Άρα θα πρέπει και οι πινακίδες και τα διάφορα αυτοκόλλητα να είναι ομαδοποιημένα και τα συστήματα πλοήγησης να είναι ομοιοποιημένα, διότι αλλιώς έχουμε μεγάλο πρόβλημα όταν ε, θέλουμε να ε, πάμε κάπου και μετά πληρώνουμε κάποιο πρόστιμο γιατί δεν ξέρουμε ε, ότι δεν έπρεπε να μπούμε και τα λοιπά. Και τελικά δεν θα έχουμε και την ελευθερία κυκλοφορίας, ιδίω για τους ε, τουρίστες. Και σε επίπεδο κοινότητας και δήμου θα πρέπει ε, να αφουγκραστούμε τις ιδέες, γιατί και στη Γερμανία υπάρχουν διάφορες τέτοιες ιδέες. Πρέπει να απευθύνουμε έκκληση στον κοινό νου ε, στη σύνεση. Ε, δεν ε, θα πρέπει να πούμε ότι όχι, το δικό μας το σύστημα είναι το καλύτερο. Χρειαζόμαστε σίγουρα απλούστευση και εναρμόνιση, όχι για το δικό μας το όφελο, για το όφελο των πολιτών και θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και σίγουρα θα πρέπει να ασχοληθεί και κατεπηγόντω η Επιτροπή Μεταφορών με αυτή την ιστορία. Έχουμε τα διάφορα προβλήματα και με, τη, με τα διόδια, τι πληρώνουν τα οχήματα, τα γιοταχή και τι πρόστιμα μπορεί να πληρώσει κάποιος που δεν ξέρει. Δεν έχω κάτι σε βάρος του συστήματος, αλλά θα πρέπει να είναι κατανοητό από όλους τους πολίτες και θα πρέπει να είναι και εναρμονισμένο. Ευχαριστώ. Μιζάουκεν. Yeah, I could agree, but... Συμφωνώ. Αλλά είναι δύσκολο. Έχουμε πολλές χώρες. Οι τουρίστες έχουν πολλές φορές προβλήματα. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, πέραν των μεθόδων του Dieselgate, το κάνανε στην Κοπενχάγη μετέφεραν τις, ε, ε τις αντλές βενζίνης μακριά από τους δρόμους και, κάνανε, και βελτιώθηκε η ποιότητα του αέρα στους δρόμους. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε άλλο. Είναι δύσκολα Υπάρχουν αιτήματα που δεν γίνονται σεβαστά. Τι συμβαίνει με την οδηγία για την ποιότητα του αέρα. Αν εγκαταλείψουμε αυτή την οδηγία θα υπάρχει ένα πρόβλημα για όλες τις χώρες. Ίσως πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο και οι τουρίστες ε, προφανώς πάντα έχουν πρόβλημα σε πολλές χώρες θα έχουν, αλλά θα μάθουν να αντιλαμβάνονται αν οι χώρες είναι ενδιαφέροντοι, ή όχι να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα. Perfecto. Pues de, después de Άκουσα την Επιτροπή, άκουσα τα μέλη της ε, Επιτροπής μας. Κρατάμε ανοιχτή την αναφορά και ζητάμε από την Επιτροπή να μας ενημερώσει αν αντιμετωπίζει τις καταγγελίες ε, που ανέφερε ο αναφέρον και μεταβιβάζουμε και στην Επιτροπή Τραν. για να ζητήσουμε τη βελτίωση της εναρμόνισης της οδηγίας. παραμένει ανοιχτό Επιτροπή Τρανς και ενημέρωση από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σημείο 13. Αναφορά 837 του 2018 του Μάρκους Μπάουμγκάρτ, Γερμανού πολίτη, για την ρήπανση του αέρα από τα αεροσκάφη. Δεν είναι παρόν ο αναφέρον. Ο κ. Φίλιπ Λέν της Επιτροπής από την ΜΟΥΒ Ευχαριστώ. Να απαντήσω στον αναφέροντα που μένει κοντά σε ένα μεγάλο αεροσκάφο και θέλει να αντιμετωπίζονται οι εκπομπέ αεροσκαφών όπω και οι εκπομπέ δίζελ από οχήματα. Ζητά ε, πανευρωπαϊκά όρια τιμών για τι εκπομπέ αεροσκαφών για να διασφαλιστεί η υγεία αυτών που μένουν κοντά στο αεροδρόμιο. Η προστασία του περιβάλλοντο είναι κομμάτι της Πολιτικής Ένωσης και περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου των μεταφορών και των αερομεταφορών. Το, η Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία είναι η πρώτη προτεραιότητα της Κομισιόν αυτής. Για τι μεταφορές και την κινητικότητα η συμφωνή μας επικεντρώνεται και στην ποιότητα του αέρα που πρέπει να βελτιωθεί κοντά στα αεροδρόμια αντιμετωπίζοντας εκπομπές και τους ρήπους από αεροσκάφη. Το 2019, τον Ιούνιο του 2019, η Επιτροπή εφάρμοσε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία την υποχρέωση να συμμορφώνεται με, τις πιο πρόσφατες, με τα πιο πρόσφατα πρότυπα μηχανών αεροσκαφών που προκύπτουν από τις οδηγίες της ΑΙΚΑΟ και μια σειρά πακέ και ένα καλάθι μέτρων για, από τη ΣΑΙΚΑΟ για τη μείωση των εκπομπών από το σύστημα αερομεταφορών. Είναι το πρώτο πρότυπο παγκόσμιες τεχνολογίες για τον κλάδο της, των αερομεταφορών με στόχο να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη αποτελεσμα... και αποτελεσματικότερη τεχνολογία στον σχεδιασμό των αεροσκαφών. Επιπλέον, το Φεβρουάριο του 2019, η ICAO ενέκρινε και, την, και πρότυπα για, τα μη πτυτικά, για, τις μη πτυτικές, για τα μη πτυτικά σωματίδια. Η ανάπτυξη των νέων αυτών προτύπων έρχεται να κλείσει ένα συνολικό πακέτο πιστοποίησης των ε, αεροσκαφών για τον ήχο, το θόρυβο των αεροσκαφών και τη, τα υπόλοιπα πρότυπα των ε, υποηχητικών αεροσκαφών εντάσσοντας, ε, που θα ενταχθούν από το 2022 στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτά τα πρότυπα δεν είναι μόνο τους, θα δουλέψει τα επόμενα έτη για να βελτιώσει τη δεσμευτικότητά τους με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού των μηχανών αεροσκαφών, τηρώντας πάντα την διεθνή νομοθεσία και την ανάγκη να υπάρξει εξισορρόπηση μεταξύ θορύβου και εκπομπών αερίων Επιπλέον η ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο λύσεων που υιοθέτησαν για την βελτίωση της διαχείρισης των αεροσκαφών στα αεροδρόμια θα επιτρέψει και την βελτίωση του περιβάλλοντος και την μείωση του θορύβου ε, που επηρεάζει τους γείτονες, ε, που, τους κατοίκους περιοχών κοντά στα αεροδρόμια. Ο κύριος Κλίνκεμπεργκ θέλει το λόγο, όχι. Ωραία. Κάποιος συνάδελφος από την Επιτροπή. No. Okay. Δεν βλέπω. Ωραία. Ο Πίτερ. Όχι, όχι, η πρόεδρος ε, ό,τι πει, συμφωνώ. Ακούσαμε την Επιτροπή, διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά και ζητούμε περαιτέρω πληροφορίες από την Επιτροπή εγγράφος για τη νέα νομοθεσία για την οποία μας μιλήσατε. Εντάξει. Ωραία. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. 14. 80, ε, αναφορά 80 του 2019 από έναν Ισπανό πολίτη για τη, της πλατφόρμα Φρένεμ La Contamination για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή Γκράουντα Καστελιών. Να καλωσορίσω τις αναφέρουσες. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας για να παρουσιάσετε το έτοιμά σας. Κατόπιν θα παρέμβει η Επιτροπή, τα μέλη της Επιτροπής και μετά θα, έχουμε, θα έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε. Καλωσορίσατε και ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε για το αίτημα που θέσατε και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με το λαό της Ταραγκόνα για την... τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η... Το θέμα μας κοντά... βρίσκεται κοντά στο Καστελιό. Είναι... Η πλατφόρμα δεν... γεννήθηκε μετά από την κόποση λόγω της έλλειψης διαφάνειας και ενημέρωσης ως προς την ε, ρήπανση στην περιοχή του Σεράγιο και Ελποερτό, κάτι που παραβιάζει την ε, σύμβαση του Άρχους για την ενημέρωση. Το Σεράγιο είναι το μεγαλύτερο ε, βιομηχανικό πολύγωνο της περιοχής της Βαλένθιας και θεωρείται ένα από τα τρία μεγαλύτερα πετροχημικά σημεία στην ε, Μεσόγειο. Δύο από αυτά βρίσκονται στα top 50, στις top 50 βιομηχανίες εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, σύμφωνα με την Κωσιόν. Ξεπερνά τους 2, τόνους, 2 ε, εκατομμύρια τόνους ανά έτος διοξιδίου του άνθρακα. Παρότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται να είναι κοντά σε πόλεις, σε λιγότερο από 2 χιλιόμετρα από πόλεις, το 67 δημιουργήθηκε, ε, χτίστηκε εκεί και ένα δηληστήριο και μετά έγιναν και, και άλλες ε, εκτάσεις. Στην Αλμασόρα, η Αλμασόρα, ένα, ένας οικισμός βρίσκεται στα 100 μέτρα. Η περιοχή ρηπαίνεται, δεν υπάρχει ενημέρωση, αλλά και πολιτικά, παρότι άλλαξε πολιτικά και το χρώμα του Δήμου και το χρώμα της περιφέρειας, δεν άλλαξαν οι συμπεριφορές. Δεν ξέρουμε ούτε τι εκπέμπεται, ούτε τι, ε, ούτε τι αναπνέουμε. Επιπλέον υπάρχει το πρόβλημα των, ε, ε της, της ε, αποθεματοποίησης των ε, ρηπαντών. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πολύ κοντά στα σπίτια βρίσκονται ε, χώροι εναπόθεσης τοξικών ουσιών. Επιπλέον βρίσκονται, βλέπουμε εξαιρετικά υψηλές, υψηλή παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων. Ζητήσαμε ε, πολλές φορές ανεξάρτητη μελέτη. Αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα το Μάιο του 2018, υποβλήθηκε έτοιμα στην Ολομέλεια και μια σειρά προτάσεων σε πολιτικό επίπεδο. Μετήχαμε σε μια σειρά συναντήσεων με το Γενικό Διευθυντή και της, της Αλλαγής του Κλίματος. Παρότι υπήρξαν κάποιες δεσμεύσεις για τη βελτίωση του ελέγχου και της διαφάνειας, οι τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις συνεχίζουν να αγνοούν τις προθεσμίες και να μην τιμούν τις υποσχέσεις τους. Ο βασικός μας στόχος είναι να προστατεύσουμε την υγεία και το περιβάλλον μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι το κλίμα είναι επίγουσα ανάγκη. Συμφωνούμε ότι είναι επίγον να θέσουμε την υγεία και το περιβάλλον πάνω από τα οικονομικά συμφέροντα. Απευθυνόμαστε στην Επιτροπή Αναφορών θεωρώντας ότι παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, έχουμε στο, στην αναφορά μας τον κατάλογο των οδηγιών που παραβιάζονται. Δεν υπάρχει μόνιμη ενημέρωση και, και στην περιοχή αυτή. Ταυτόχρονα δεν υπάρχουν ανεξάρτητες και πλήρεις μελέτες για την ποιότητα του αέρα που λαμβάνουν υπόψη την εγκύτητα αστικού, του αστικού χώρου παρέχοντας ρεαλιστικά στοιχεία βάσει των οποίων να μπορέσουν να υιοθετηθούν διορθωτικά μέτρα. Για όλου αυτού του λόγου, ερχόμαστε εδώ με πέντε συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτον, η Επιτροπή Αναφορών να απευθυνθεί γραπτό προ την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, εκφράζοντα την ανησυχία τη και ζητώντα να δοθούν στου πολίτε και στην πέτεια ανεξάρτητε πληροφορίε που είναι αναγκαίε για να γνωρίζουμε τι αέρα αναπνέουμε. Δηλαδή, να ασκηθεί πίεση ούτω ώστε να τηρηθούν οι διατάξεις της Σύμβασης του Άρχους για τη διαφάνεια και τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, καθώς και ολόκληρη η εφαρμοστέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεύτερον, η Επιτροπή αυτή να ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να τηρήσουν τις ελάχιστες υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τις ενώσεις πολιτών και που εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια του Δήμου, μόνιμους σταθμούς μετρήσεων στα βασικά σημεία κλειδιά για την ποιότητα του αέρα να αναζητηθούν επίγουσες λύσεις για να σταματήσουν να περιορίζονται η, η εκπομπή ελεύθερων σωματιδίων στην περιοχή του λιμανιού με σωματίδια σκόνης και ταυτόχρονα να αποσταλεί αντιπροσωπεία βουλευτών της Επιτροπής Αναφορών για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να εξετάσουν διεξοδικότερα το ζήτημα. Και ζητούμε η Επιτροπή και η αναφορά να παραμείνει βεβαίως ανοιχτή και να παραμείνουν ε, τα αιτήματα ενημέρωσης μέχρι ότου δοθεί λύση στο πρόβλημα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Λουθία Μπερνάλ από την ΕΜΒΗ. Thank you, Chair. Here. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μου δίνετε το λόγο αλλά θα τα ναι. πω ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες ε, για την ε, παρουσίαση των γεγονότων από την πλατφόρμα Φρένε Μπλακών Ταμιναθιό. Θέλω να πω ότι σε ό,τι αφορά την ρήπανση και την ατμοσφαιρική ιδιαίτερα, ε, είναι πολύ σημαντικές περιβαλλικές προτεραιότητες για την Κομισιόν λόγω των σοβαρών επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία, τα οικοσυστήματα αλλά και την οικονομία των κρατών μελών. Ως ήδη ενημερώθηκε από τον Αύγουστο του 2019 η Επιτροπή σας από την Κομισιόν, η ανάλυση των σχεσμών των αναφερόντων δεν επέτρεψε παρόλα αυτά να φανεί ότι υπάρχει ε, μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την Ισπανία. Παρ' όλα αυτά σημειώσαμε τις πληροφορίες που έδωσαν στην Επιτροπή σας οι αναφέροντες και όταν ανα, ε, λύσουμε τις πληροφορίες θα σας στείλουμε γραπτό στα σχόλιά μας και τα συμπεράσματά μας. Δεύτερον, η οδηγία για τις εκπομπές, τις βιομηχανικές, είναι το βασικό εργαλείο της Ένωσης για τη ρύθμιση των ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις μονάδες περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής οδηγίας ε, θα πρέπει να έχουν ε, άδειε που περιλαμβάνουν ωραίες τιμές εκπομπών για εκπομπές ρήπου στην ατμόσφαιρα, στο νερό και στο έδαφος, αλλά να περιλαμβάνουν και τις απαιτούμενες διατάξεις για τον έλεγχο των εκπομπών. Όλα αυτά θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Η οδηγία επομένω θεσπίζει κανόνες για την πρόσβαση σε πληροφορίες και για τη συμμετοχή της κοινή γνώμη και εγγυάται στου διαβεβαιωμένους πρόσβαση στη δικαιοσύνη εφόσον δεν τηρούνται οι δεσμεύσει και υποχρεώσει ε, Η οδηγία για την ε, ποιότητα, ε, η πρόεδρος, λίγο πιο αργά παρακαλώ, για να μπορούν να σας παρακολουθούν οι διερμηνείς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έλεγα ότι οδηγίε για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ορίζουν ορικέ τιμέ για τρει ε, ατμοσφαιρικού ρήπου που δεν πρέπει να ε, υπερβαίνονται για την προστασία τη δρόμων υγεία και την προστασία του περιβάλλοντο. Ε, παρακολουθούμε και του σύνοικη ε, την εφαρμογή των οδηγιών. Αν υπάρξει παραβίαση και συστηματική, θα παρακολουθεί το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με διαδικασίες επί παραβάση ε, σε βάρος ε, των ε, εκάστοτε κρατών μελών. Και για την περίπτωση της Ισπανίας έγιναν διαδικασίες επί παραβάση επειδή έχουν παραβιαστεί οι οριακές τιμές για το PM10 και για το διοξίδιο του αζότου σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις και συγκεκριμένες περιοχές. Ό,τι αφορά το διοξίδιο του αζότου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης να προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί δεν τηρεί τις σχετικές ε, διατάξεις η Ισπανία. Πρέπει να πούμε όμως ότι ανάλυσε τις δύο τελευταίες εκθέσεις Κομισιόν για την ποιότητα του αέρα, εκθέσεις που έστειλαν οι Ισπανικές Αρχές, σε ό,τι αφορά το 1050 Καστεγιώνα σε μια περιοχή που βρίσκεται το Σεράγιο. Εκεί δεν υπήρξε υπέρβαση καμία οριακή ε, τιμή σε σχέση με αυτές ε, που θεσπίζει η οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Ούτε το 2017 ούτε το 2018. καλούνται τα κράτη-μέλη να τηρούν τι ενδεικτικέ τιμέ για την ποιότητα του αέρα όπω προβλέπονται από την ε, Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία. Αλλά οι μόνε ορκέ τιμέ που υποχρεωτικά πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη είναι αυτέ που προβλέπονται στι οδηγίε που προανέφερα. Τέλο. Η ζώνη ποιότητα ε, το ατμοσφαιρικού αέρα λαμβάνει υπόψη τις, τις τιμές του παραρτήματος της οδηγίας. Άρα για τη σωστή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει και η δεματοληψία να γίνεται σωστά σημεία, αλλά αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μέλων, όπως και για όλα τα άλλα. Ζητούμε λοιπόν να ενημερωθούν ε, αρχές από τους αναφέροντες για τις πληροφορίες που έχουν και να στραφούν, αν αυτό καταστεί αναγκαίο, στο Εθνικό Δικαστικό Σύστημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιο από την Κομισιόν που θα θέλει το λόγο από την Επιτροπή μας μάλλον που θα ήθελε το λόγο. Yes. Something... Κυρία okay. ίσως να είμαι κουρασμένη. Κάτι με ενοχλεί όμως. Δεν γίνεται σεβαστή η σύμβαση του άρχους. Αν δεν γίνεται σεβαστή, οι αναφέροντες και οι πολίτες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα πραγματικά στοιχεία. Γι' αυτό ίσως είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα απαντώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέτε ότι δεν υπάρχει παραβίαση ενωσιακού δικαίου. Έχουμε και οδηγία για βιομηχανικές εκπομπές. Γίνεται σεβαστή. Άκουσα την αναφέρουσα. Τις αναφέρουσες είπαν και ότι είναι απαράδεκτη κατάσταση από πλευρά ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα. Να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, λέω. Να εξετάσουμε ποιε οδηγίε έχουν παραβιαστεί. Φαίνεται επίγον το θέμα για δημόσια υγεία και περιβάλλον. Ίσως να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και να μην έχει παραβιαστεί τίποτα, αλλά δεν μου φαίνεται ότι είναι έτσι. Ευχαριστώ. Ah, Ευχαριστώ πολύ, Πέτερ Γιάρ. Δύο προβλήματα βλέπω. Το πρώτο, η απάντηση της Κομισιόν ε, ήταν κάπως διαφοροποιημένη. Δεν είπε ότι είναι όλα καλά. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια διαβήματα ε, στην Ισπανική ε, κυβέρνηση. Τέλο πάντων να υπάρξει ένα είδος διαλόγου. Τώρα το δεύτερο, διαφάνεια. Είχαμε πάει σε μια επίσκεψη διερευνητική στην Ιταλία που ουσιαστικά περί το ίδιο επρόκειτο. Είχαν πει ότι τα πράγματα είναι εντάξει αρχές και οι πολίτες είχαν πει ότι δεν είναι εντάξει τα πράγματα. Και τελικά ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και το πώς αισθάνεται ο κόσμος. Ε, δεν υπάρχει οικοδόμηση εμπιστοσύνη κατά αυτόν τον τρόπο οι αναφέροντες. Νομίζω ότι έχουν δίκιο όταν λένε ότι θέλουμε να ξέρουμε τι μας ε, μετράτε εδώ, τι, τι μετράτε, πώς θα μετράτε. Πρέπει αυτά να γίνονται με διαφανή τρόπο. Γιατί αν δεν υπάρξει διαφάνεια, τότε υπάρχει ε, έλλειψη εμπιστοσύνης ε. Επομένως, ναι, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και η Κομισιόν θα πρέπει νομίζω να καθίσει να πραγματευτεί με τις Ισπανικές Αρχές για ορισμένα πράγματα. Και πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος των αρχών με τους πολίτες, ε, να τους λένε ακριβώς ε, περί τίνος πρόκειται, τι μετράνε ακριβώς, γιατί αλλιώς δεν οικοδομείται εμπιστοσύνη, όπως είπα. Όταν δεν δημοσιοποιείται κάτι, δημιουργούνται πάρα πολλές έτσι, επιφυλάξεις ε, και υποψίες. Έτσι είναι η ζωή. Άρα πρέπει να συζητούνται αυτά ανοιχτά, με διαφάνεια. Και όταν υπάρχει διαφάνεια, έπειτα θα συζητήσουμε κατά πόσον το πρόβλημα λύθηκε ή όχι. Αλλά πρώτα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Ευχαριστώ. η ε, κυρία Βιανουέβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να ευχαριστώ την ε, πλατφόρμα αυτή κατά της ρήπανση που έφερε αυτή την αναφορά στην Επιτροπή μας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μας προειδοποιεί πολύ θάνατοι ε, από την ε, ατμοσφαιρική ρήπανση, πάνω από 7 εκατομμύρια στον κόσμο, 10.000 στην Ισπανία από, πεθαίνουν από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Ακούσαμε την πλατφόρμα για το Σεράγιο, είναι μια βιομηχανική περιοχή στη Βαλένθια που υπάρχουν πολλές πετροχημικές ενεργειακές επιχειρήσεις και είναι ε, ένας από τους τρεις μεγαλύτερους πετροχημικούς κόμπους στη Μεσόγειο. Χιλιάδες κάτοικοι από το Αλμασόρα, από το Καστεγιόν ε, έχουν ε, πολλά προβλήματα αναπνευστικά, υγείας, λόγω της εισπνοής όλων αυτών ε, των σωματιδίων ε, και των ρήπων που εκπέμπονται από τις δραστηριότητες εκεί και από τη σκόνη που αιωρείται. Επίσης, οι περιφερειακές αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε κάποια λύση. Ο αγώνα κατά τη κλιματική αλλαγή ο αγώνα και κατά αυτών που, έχουν, ε, έχουν, που ευθύνονται για αυτά τα υψηλά επίπεδα ρήπανση. Δεν μπορούμε να βάζουμε τα εμπορικά συμφέροντα πάνω από τη ζωή και την υγεία του κόσμου. Θέλω λοιπόν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να υπάρξει επαφή με τις αρχές, τις τοπικές, περιφερειακές, να καταδειχθεί η ανησυχία μας και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Στηρίζω επίσης να έχουμε την απαραίτητη μέτρηση, τα απαραίτητα όργανα μέτρησης εκεί που πρέπει, ώστε επίσης ε, να μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες και για το VTX ιδίω. Να υπάρχουν κατάλληλοι μετρητέ, να μπορούν να στέλνουν οι πολίτε ε, δείγματα και να παίρνουν ε, απαντήσει. Να ζητήσω λοιπόν να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να ζητήσουμε εξηγήσει ε, από τι τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Έχετε δύο λεπτά τώρα οι αναφέρουσε. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε μελέτη, ανεξάρτητη μελέτη για την ποιότητα του αέρα στην περιοχή του Σεράγιο. Άρα δεν γνωρίζουμε αν ε, υπάρχουν ή όχι αυτοί οι 13 ρηπαντές. Δεν υπάρχει επίσης σταθμός, σταθερός σταθμός μέτρησης μέσα στον οικισμό. Ο μόνος που έχουμε βρίσκεται στην άλλη πλευρά του χωριού. Άρα οι εκπομπές το κατά πόσο ξεπερνιούνται ή όχι οι εκπομπές είναι κάτι το αβέβαιο. Όπως αναφέρθηκε εδώ, η έλλειψη ενημέρωσης, η ελλειψη ενημέρωση, διαφάνειας δημιουργούν μεγάλες ανησυχίες. Γι' αυτό ζητούμε από την Επιτροπή Αναφορών να κρατήσει ανοιχτή την αναφορά αυτή και να ζητήσει πληροφορίες, περισσότερες από αυτές που αναφέρονται και από τις επιχειρήσεις της ίδιας. Όταν λέμε ότι παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ε, εννοούμε ότι κάτι που δεν έγινε καλά μπορεί να ήταν η εφαρμογή, η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία. Ξέρετε ότι τις οδηγίες τις εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Η περιφερειακη νομοθεσια ξερετε οτι τις οδηγιες μεριμνά για την τήρησή τους. Γι' αυτό θέλουμε να στραφούμε προς την Επιτροπή για να ζητήσουμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά έως ότου έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το αέρα που αναπνέουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Έχοντας ακούσει την Επιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής μας προτείνω να μην ανοιχτεί η αναφορά. Δεύτερον, να συνεχίσουμε να ζητούμε από την Κομισιόν όλες τις ε, πληροφορίες, διότι όπως εξήγησε η Κομισιόν στην περιοχή του Καστελιών το 2018-19 δεν ξεπερνιόντουσαν οι παραμετροί, αλλά όπως αναφέρθηκε, ε, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Επιτροπής, ήταν, θα υπάρξει μια νέα ενημέρωση για την περίπτωση αυτή. Ζητούμε λοιπόν από την Κομισιό να μας ενημερώσει για το τι κάνουν ώστε να αξιολογήσουν την κατάσταση. Τρίτη απόφαση να στείλουμε στις Ισπανικές Αρχές ιδίως στο στο Υπουργείο για την Οικολογική Μετάβαση και την, ε, το Υπουργείο Γεωργίας Ανάπτυξης ε, Κλιματικής Αλλαγής και Οικολογικής Μεταφοράς της ε, Περιφέρειας της Βαλένσια. Αυτό λοιπόν κάνουμε και αφήνουμε ανοιχτή την Επιτροπή. Τώρα, το πέμπτο σημείο που ανέφερα, το τέταρτο σημείο που ανέφεραν οι αναφέρουσες, να πάει μια αντιπροσωπεία ε, βουλευτών είναι αρμοδιότητα των συντονιστών κάθε, που περιλαμβάνει τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων. Αυτό αποφασίζεται μία φορά το χρόνο, άρα τον Οκτώβριο, τον Οκτώβριο του 19 αποφασίσαμε τις αποστολές για το 20. Σας το λέω, που, να ξέρετε πώς λειτουργεί το θέμα των αποστολών. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, γιατί πρέπει να σταματήσουμε στις 6.30. Έχουμε και άλλες αναφορές. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή Αναφορών είναι η γέφυρα μεταξύ των πολιτών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά πράγματα επιτυγχάνουμε εδώ για να φέρουμε πιο κοντά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους πολίτες της Ένωσης. Συνεχίζουμε. Σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης. 943 του 2008. Αναφορά Γερμανού πολίτη για την ερμηνεία και εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης ε, της ατμοσφαιρικής ρήπανσης στη Γερμανία και τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Δεν είναι εδώ ο αναφέρον. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ένβη, ο κύριος Κρίνκεμπεργκ. Ευχαριστώ. Um, Να πω περί τίνος πρόκειται. Ζητάει ο αναφέρον περιορισμούς οχημάτων, κυρίως διζελοκίνητων, σε πόλεις της Ευρωπαϊκής Ενώσης λόγω ρήπανσης. Και ρωτάει γιατί αυτοί οι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εναρμονισμένα, γιατί υπάρχουν διαφοροποίησεις μεταξύ Γερμανίας κυρίως και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνηση. Αντίθετα με αυτά που αναφέρεται στην αναφορά, έχουμε νόμους για χαμηλές εκπομπές σε αρκετές χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να μειωθεί εκπομπή ρηπαντών από την κυκλοφορία. Σε γραπτή απάντηση δώσαμε ένα σύνδεσμο στο διαδίκτυο που μπορεί κανείς να τα δει όλα αυτά τα στοιχεία. Τι έχει γίνει πού και κάτι άλλο. Προς διευκρίνηση. Η απόφαση θέσπιση ορίων χαμηλών για εκπομπέ δεν είναι κάτι που λαμβάνεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε στην οδηγία για τον περιβαλλοντικό αέρα, καθορίζονται οριακέ τιμέ για συγκεντρώσει ρηπαντών και τα πρότυπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η υποχρέωση για τα κάτι μέλη υπάρχει για αποτελέσματα. Δεν υπάρχει υποχρέωση για τρόπους επίτευξης των αποτελεσμάτων. Οι τρόποι που χρησιμοποιούνται δεν προκαθορίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. και αν λαμβάνονται μέτρα για αποφυγή ρήπανσης από κυκλοφορία, σημαίνει ότι η οδηγία δεν δίνει δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή συγκεκριμένων μέτρων που θα επιβάλλουν η τοπική αυτοδιοίκηση ή οι εθνικές αρχές. για τυχόν περιορισμούς και άλλα μέτρα. Τούτων λεχθέντων, ποιο είναι το γενικό πλαίσιο και η λειτουργία της νομοθεσίας. Προσπαθώ να περιγράψω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει υπερβάσει συγκεντρώσεων στη Γερμανία στον αφορά του ρηπαντέ και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση για υπερβάσει ετήσιου ορίου ε, οξυδίου του αζότου, ε, διοξιδίου του αζότου στην ε, Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρεμβαίνει και δεν μπορεί άμεσα να παρέμβει βάσει των οδηγιών για να επιβάλλει μέτρα όπως ζώνες για χαμηλές εκπομπές ή άλλους περιορισμούς, πώς θεσπίζονται τα μέτρα βάσει πρίων κριτηρίων, όμως υπερβάσεις ρηπαντών και οριακών τιμών τις αντιμετωπίζουμε μέσω διαδικασιών επί παραβάση και έχουμε κάνει μια τέτοια διαδικασία, έχουν ξεκινήσει κατά της Γερμανίας. Ευχαριστώ. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιάρ. Ναι, ευχαριστώ. Η απάντηση Κομισιόν. Σωστή ήταν, παρόλα αυτά, εγώ θα ήθελα να μείνει ανοιχτή αναφορά. Σε σχέση και με το σημείο 11, η εναρμόνιση ε, των μέτρων για την ατμοσφαιρική ρήπανση. Σωστά τα είπατε ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την τήρηση των οριακών τιμών, και ότι θα πρέπει να ληφθούν σε περιφερειακό επίπεδο μέτρα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε δεκτή μεταχείριση των πολιτών. Θα πρέπει δηλαδή, να υπάρχει σαφής γνώση και κατανόηση, θα πρέπει να είναι ευληπτά τα μέτρα και τρίτον να ενημερώνονται οι πολίτες. Λέω, να μείνει ανοιχτή αναφορά και να την ε, στείλουμε και στην Επιτροπή Μεταφορών. Όχι ότι έχω κάτι σε βάρος των μέτρων, απλά τελικά ε, υπάρχει μεν ελευθερία είτε δεν υπάρχει. Ε, γιατί αν εγώ πάω στην Γαλλία πάντα φοβούμαι ε, και κοιτάω δεξιά και αριστερά πώς κάνω κάτι λάθος ε, και πληρώσω πρόστιμο μετά. Οπότε νομίζω ότι από τη μία υπάρχει το δικαίωμα ελευθερίας μετακίνησης για τους Ευρωπαίους πολίτες αλλά και η ανάγκη εναρμόνισης ε, για να βελτιωθεί η ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα. Εγώ λέω να μείνει ανοιχτή αναφορά και να συζητηθεί και από την Επιτροπή Μεταφορών το γιατί τελικά έχω όλα αυτά τα, ε, αυτοκόλλητα για την ατμοσφαιρική ρήπανση και δεν ξέρω εγώ για τα τέλη και το ένα και το άλλο, αλλά όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο αναγκαιώνται την ε, ελευθερία μετακίνησης. Ε, πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, κάποιος απλός κανόνας. Όποιος οδηγεί πληρώνει. Κάτι απλό να μην την πατάμε αν νομίζουμε ότι είμαστε, ξέρω εγώ, σε έναν τοπικό δρόμο και έχουμε βρεθεί σε αυτοκινητόδρομο και μετά πληρώνουμε πρόστιμα. Επειδή θέλαμε να επισκεφθούμε την όμορφη Ευρώπη αλλά δεν ε, ξέραμε τι ισχύει, και δεν ξέρω επίσης εάν ε, μπορεί κανείς ε, να πληρώνει ηλεκτρονικά εφόσον γνωρίζει το σύστημα και αυτούς, αυτά τα τέλη και όχι να πληρώνει μόνο τους φόρους και τα πρόστιμα, μάλλον τα πρόστιμα. κυρία Όκεν, να πω στον Πίτερ, ναι. Και εσείς έχετε δικαίωμα να πεθάνετε νωρίτερα από τη ρήπανση του ατμοσφαιρικού αέρα. Δεν κάνω διάκριση. 800.000 άνθρωποι πεθαίνουν πρώιμα λόγω μολυσμένου αέρα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε διάκριση εδώ λοιπόν. Πρέπει να αναρμονίσουμε και πού θα γίνουν οι μετρήσεις. Όπως πριν που συζητάγαμε την άλλη αναφορά. Και όπως ανέφερα και εγώ την Κοπενχάγη, που μετακίνησαν την μέτρηση για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και η ποιότητα του αέρα. Ίσως πρέπει να επιμένουμε να υπάρχει σωστός τρόπος μέτρησης. Μέσω των αναφορών δημιουργείται εντύπωση ότι γίνονται πολλά κόλπα. Και πρέπει να είμαστε πολύ πιο σκληροί. Ακόμα και εσύ, Πίτερ, πρέπει να επιβιώσεις. just a small... Λοιπόν, σχόλιο για τον σφαιρική ρήπανση δεν είναι πρόβλημα μιας χώρας και μόνο, είναι διασυνοριακό πρόβλημα. Αισθητό σε όλους και σπαράγεται αλλού. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους. Χρειάζεται και άλλη δουλειά για εναρμόνιση. Άρα, η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή. Thank you very much. Okay. So our proposal is to maintain... Άρα η πρόταση είναι να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για την ε, όλη εξέλιξη της διαδικασίας. Εντάξει, ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 9, συνεδρίαση συντονιστών και στις 10, συνεδρίαση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.